Bene, benvenuti a tutti, possiamo iniziare il... Μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με την μήνυα κράση που έχουμε, αλλά βέβαια αφού εγκρίνουμε την μερίσια διάταξη. Αν συμφωνείτε, εγκρίνει τη μερίσια διάταξη. Για τις ανακοινώσεις, η μόνη ανακοίνωση που πρέπει να σας κάνω, αλλά μπορώ να το κάνουμε για να έρθουν και οι συνάδελφοι αργότερα, είναι ότι σήμερα, σε αυτή την αίθουσα, ε, έχουμε 12 καμπίνες για διερμηνία. Επομένως, έχουμε μόνο 12 γλώσσες στη διάθεσή μας με βάση την σύνθεση της Επιτροπής μας. Μπορούμε τώρα να περάσουμε άμεσα σε αυτή την μίνι ακρόαση για τις προοπτικές της βιομηχανίας και της έρευνας με βάση το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Οι προοπτικέ του Γενικού Κανονισμού την προστασία των δεδομένων όσον αφορά την βιομηχανία και την έρευνα. Για τη συζήτηση αυτού του θέματος έχουμε μέχρι τις 5 και 4 το πολύ και το πρώτο κομμάτι θα το αφιερώσουμε στις παρεμβάσεις των συναδέλφων και μετά θα ακούσουμε τους δύο ε, φιλοξενούμενού μας, τους δύο προσκεκλημένους μας. Για πέντε λεπτά θα δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο Κέλλη, που είναι και η εισηγητής για να μιλήσει εξ ονόματος της ε, Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ πέντε λεπτά. Αλλά καταρχάς, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι είναι τιμή για μένα που ξεκινάω εγώ ε, τις παρεμβάσεις για, αυτόν τον, ε, για αυτή τη συζήτηση για τις προοπτικές του Γενικού Οργανισμού για την των Δεδομένων όσον αφορά τη βιομηχανία και την έρευνα. Ε, σαν εισηγητής ε, συνεισέβαλα στην δημιουργία αυτής της ακρόασης γιατί πιστεύω ότι οι προοπτικές βοηθάνε ιδιαίτερα να, βελτιώσουμε την ε, καθημερινότητά μας, το περιβάλλον της πόλης κτλ. και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Ε, είναι μια, ένας για, για την επίτευξη των στόχων για την Ευρώπη του 2020 και ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε καινοτομίες. Όμως χρειάζεται ένα στέρεο νομικό πλαίσιο που να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, γι' αυτό είμαστε εδώ ε, σήμερα. Δεν πρόκειται να σας καθυστερήσω. Καλό είναι να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες που θα μας δώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά αυτόν τον κανονισμό έτσι ώστε να μας δώσουν τα φώτα τους για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές και αλλαγές έτσι ώστε να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο. Ε, χαίρομαι γιατί η πρόοδος γίνεται, εμφανίζεται ταχύτατα. Ε, είχαμε πολλές συναντήσεις ε, με εκπροσώπους της, του επιχειρηματικού κόσμου, των καταναλωτών. Όσοι θέλανε να μας συναντήσουν, τους συναντήσαμε. Και Είχαμε και πολλές συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές, με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι ο, πρόεδρο, ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας ε, μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι θα ήθελε να θέσει σαν υψηλή προτεραιότητα την προστασία των δεδομένων όσον αφορά την βιομηχανία και την έρευνα. Δηλαδή αυτό το θέμα θα έχει μεγάλη προτεραιότητα στην ατζέντα της Ιρλανδικής Προεδρίας, θα συζητηθεί από την αρχή και θα προχωρήσουμε σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και ελπίζω ότι το επόμενο εξάμεινο στην Ιρλανδική Προεδρία θα προχωρήσουμε γρήγορα και να ε, ολοκληρωθεί το όλο θέμα κατά διάρκεια της Λιθουανικής και μετά της Ελληνικής Προεδρίας που θα ακολουθήσουν. Διότι είναι σημαντικό ε, σε αυτή την ε, εντολή, σε αυτή την ε, θητεία τέλος πάντων, να, σε αυτές τις θητείες να ολοκληρωθεί Γι' αυτό καλό είναι να ακούμε τις απόψεις των ενδιαφερομένων και να εξετάζουμε τις συνέπειες των προτάσεων στο γενικότερο πλαίσιο των συνεπειών στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, γιατί υπάρχουν διαφορές. Γι' ανάμεσα στους κλάδους. Γι' αυτό θα πρέπει να, το, να λάβουμε υπόψη μας το σύνολο των συνεπειών και να προσαρμόσουμε ανάλογα τις ε, προτάσεις μας. Γι' αυτό ακριβώς ε, η σημερινή συνεδρίαση είναι υψής της σημασίας θα έλεγα. Και με αυτές τις προκαταρκτικές ε, παρατηρήσεις δίνω το λόγο στον Πρόεδρο και περιμένω να ακούσω με υπομονησία την παρέμβαση. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Κέλλη Ξεκινάω αμέσως. Α, εδώ είναι ο εισηγητής μας, εντάξει. Δεν βλέπω πάρα πολύ καλά από εδώ. Μου είπαν ότι δεν είσαστε εδώ, αλλά τελικά ήσασταν. Ο κύριος Άλμπρεχτ, ο εκπρόσωπος των φιλελευθέρων έχει και... της Επιτροπής ε, Ελευθεριών, έχει και αυτός ε, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τέλο πάντων, δεν με αναγνωρίσατε, αλλά έχει το καρτελάκι το όνομά μου εδώ μπροστά, νομίζω. Τέλο πάντων, σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για αυτή την μήνυα ακρόαση. Χαίρομαι πολύ που έχουμε πλέον και κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που θα συζητήσουμε, τα ευφύ δίκτυα, την έρευνα, πολύ σημαντικά σημεία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το θέμα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ σε όλη την ακρόαση, αλλά θα ήθελα στην αρχή να εκφράσω κάποιες απόψεις και για την κατάσταση πρώτη των εργασιών μας στην Επιτροπή Λίμπη. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε βέβαια πρώτα απ' όλα τα Χριστούγεννα, αλλά θα έχουμε δύο εκθέσεις για την, ε, το πακέτο μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων στις 10 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τις, ε, τις διακοπές δηλαδή και θα έχουμε και την έκθεση για τον κανονισμό και την έκθεση για την οδηγία. Εν συνεχεία, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, θα υπάρξει δυνατότητα για τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να καταθέσουν τροπολογίες στην έκθεση και βέβαια θα πρέπει να καταλήξουμε και σε συμβιβασμούς. Και αυτό να το κάνουμε τάχιστα για να μπορέσουμε να έχουμε ψηφίσει πριν το καλοκαίρι και να ξεκινήσουν έτσι οι διαπραγματεύσεις με την Ιρλανδική Προεδρία, όπως είπε πολύ σωστά ο Σον Κέλλη. Αυτός είναι ο στόχος μας, είναι προτεραιότητα το θέμα και είναι σημαντικό να είναι και στο Συμβούλιο ταχεία διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να ξεκινήσουμε μετά το καλοκαίρι τις διαπραγματεύσεις και να ολοκληρώσουμε αυτή την νομοθετική μεταρρύθμιση πριν τις ευρωεκλογέ. διότι φαντάζομαι ότι αν δεν το πετύχουμε αυτό, με το νέο κοινοβούλιο που θα έχει συγκροτηθεί και με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Και ίσως χρειαστεί να ξαναξεκινήσουμε πολλά πράγματα από το μηδέν. Έχει ήδη γίνει όμως πάρα πολλή δουλειά φέτος, όλη τη χρονιά πραγματικά είχαμε πολλές συναντήσεις, και συνεδριάσεις και με τον συντάκτη και με όλους τους υπόλοιπους. Θέλουμε λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε οι επιτροπές. Είναι πολύ καλό. Τώρα να σας μιλήσω λίγο για την όλη προσέγγιση. Είναι σημαντικό να λέμε και να τονίζουμε ότι δεν θέλουμε να αλλάξει άρδινο τρόπος ε, κατάρτιση νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Η σημαντικότερη στόχη μας είναι καλύτερη εναρμόνιση, άρα και καλύτερη εφαρμογή των κανόνων που έχουμε ήδη στην οδηγία 9546, διότι υπάρχουν στα κράτη-μέλη διαφορετική τρόποι εφαρμογή και υπάρχει και έλλειψη ε, στην επιβολή της νομοθεσίας, το έχουμε δει επί σειρά ετών. Η θέση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι ξεκάθαρη ήταν ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση, γι' αυτό και προτείνουμε έναν κανονισμό. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη εφαρμογή, αλλά θέλουμε και επιβολή κυρώσεων. Και επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε και τα μεμονωμένα δικαιώματα. Έτσι ώστε όλοι στην Ευρώπη γνωρίζουν ποια είναι τα μεμονωμένα δικαιώματα που εφαρμόζονται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Κάτι άλλο σημαντικό όμως ε, είναι ο στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, οι αρχές, οι πολίτες, οι πελάτες να μπορούν να βασίζονται στους κανόνες, να έχουν ασφάλεια δικαίου. Αυτό να ισχύει σε όλη την Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, από όπου και αν προέρχονται αυτές. Αν επεξεργάζονται δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών ή πελατών, θα πρέπει να διέπονται από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία αυτή, είναι και θέμα προστασίας και διασφάλισης ε, του ίδιου επίπεδου ανταγωνισμού. Έχουμε τους κανόνες ανταγωνισμού για επίσης για την προστασία των δεδομένων και νομίζω θα ήταν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους να συζητούμε και για τον αντίκτυπο στην αγορά εν γέννη πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη το τεράστιο λοιπόν όφελος και πλονέκτημα που θα δώσει στον τομέα των επιχειρήσεων αυτή η νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή έχουμε οδηγία. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν οι διατάξεις σωστά. Δεν θέλουμε να φορτώσουμε επιπλέον τις επιχειρήσεις, δεν θέλουμε περαιτέρω κανόνες περαιτέρω άχθος, γιατί αν πούμε κάτι τέτοιο, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Τέλος πάντων πρέπει να κάνουμε ξεκάθα πού είναι τα ισχυρά σημεία, πού είναι δυναμίες και νομίζω ότι και από την αμήνευτη ακρόαση θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα. Θα συμφωνήσουμε δηλαδή για τους κανόνες που ισχύουν ήδη και για αυτούς που θα προταθούν μέσω του κανονισμού. Επίσης, όταν ε, στην ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα υποβάλουμε αυτές τις εκθέσεις στις 10 Ιανουαρίου. Θα έχουμε λάβει υπόψη μας ε, πάρα πολλές απόψεις από τους ενδιαφερόμενους ε, φορείς και επίσης από τους σκιώδεις, από τις επιτροπές. Όλα αυτά θα τα έχουμε συλλέξει ένα σχέδιο κειμένου και θα ήθελα να μελετήσετε αυτό το κείμενο. Θα είναι έτοιμο αρχές Ιανουαρίου. Νομίζω ότι θα είναι ένα νέο έγγραφο εργασίας το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και ελπίζω του χρόνου να καταλήξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Άλμπρεχτ. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα, η ακρόαση θα χωριστεί σε δύο ε, κομμάτια. Το πρώτο θα αφορά την έρευνα και το δεύτερο την βιομηχανία. Για 8 λεπτά τον λόγο έχει η Jessica uh, first of all, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ που ε, με καλέσατε. Είναι τιμή ε, για μένα. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω καταρχάς ποιοι είμαστε για να γνωρίζετε ποιο είναι το πλαίσιο. Η SEDC ε, είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσπαθεί να ασχοληθεί ε, με ε, όλες τις ε, βιομηχανίες, με όλες τις επιχειρήσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη και ασχολείται με την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στην ενεργειακή αγορά μέσω feedback, μέσω δυναμικής τιμολόγησης καλύπτει τέλος πάντων ε, τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη διασφάλιση μέγιστης αποτελεσματικότητας ε, της ενεργειακής αγοράς, όπως επίσης και τη μεγιστοποίηση των, του ωφέλους για τους καταναλωτές. Θα ήθελα καταρχάς να σας μιλήσω για την εκτίμησή μας για την αναγνώριση του κυρίου Κέλλη ότι η προστασία των δεδομένων πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλες πολιτικές ε, και άλλες προτεραιότητες πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο και πολύ ε, δραματικό παράδειγμα στον τομέα δηλαδή της ενεργειακής αποτελεσματικότητας θα αναφερθώ και ειδικότερα στον τομέα του informative billing, της ε, ενημερωμένης τιμολόγησης αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι ότι μπορεί η προστασία δεδομένων ε, να απειλεί τη δυνατότητα των ε, επιχειρήσεων για την παροχή ενημέρωσης. Να σας πω δηλαδή τι εννοώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το feedback, ε, οι πληροφορίες σημαίνουν ε, κάποιου είδους ε, εκπαίδευση. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση του πώς οι καθημερινές μας δραστηριότητες επηρεάζουν ε, το πόσο στοιχίζουν οι λογαριασμοί μας και τι ακριβώς σημαίνουν αυτοί οι λογαριασμοί σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση. Η συμπεριφορά μας και, ο, και ο, η ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουμε δεν ε, διασταυρώνονται ποτέ. Δηλαδή δεν, δια, δεν διαπιστώνουμε πόσο πολύ ε, ενέργεια καταναλώνουμε. Για παράδειγμα, ο ζεστός ε, καφές που μόλις γίνεται ε, στο φλιτζάνι σας χρειάζεται ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός λοιπόν που καταναλώνει αυτός ο ζεστός καφές και η συμπεριφορά μας ζητώντας ζεστό καφέ δεν διασταυρώνονται. Εμείς αυτό, το feedback ακριβώς συνδυάζει τις δράσεις με ε, τα αποτέλεσμα και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε υπεύθυνες επιλογές, υπεύθυνες επιλογές που επίσης ε, είναι υποφελείς για μας. Ένας ε, πολύ βασικός τρόπος είναι μέσω, για παράδειγμα, ε, ενημερωμένους λογαριασμούς, οι περισσότεροι δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται ένας λογαριασμός σας, ε, δεν γνωρίζετε πόσο πληρώνετε το μήνα και δεν ξέρετε και τι ακριβώς, σε τι ακριβώς ε, αντιστοιχεί αυτό. τι χρησιμοποιούμε, τι καταναλώνουμε περισσότερο. Καταναλώνουμε 40-50% του ηλεκτρισμού μας το βράδυ, ε, αν έχουμε το σχετικό πρόγραμμα. Μπορούμε, μπορούν δηλαδή οι εταιρείε να δώσουν τι πληροφορίε αυτές στου καταναλωτέ και η ανταπόκριση, και το λέω ε, αυτό ε, έχοντας ρωτήσει 450.000 καταναλωτές, ε, η μείωση της κατανάλωσης όσων συμμετείχαν σε προγράμματα ενεργειακής ε, κατανάλωσης είναι πάρα πολύ σημαντική και το λέω αυτό σε σχέση μόνο με το λογαριασμό, κάτι το οποίο προσπαθούμε μέσω των εφιών ε, ε, μετρητών μας να προσμετρήσουμε. Ορισμένα πράγματα θα ήθελα να πω για να είναι πιο αποτελεσματική αυτή η τιμολόγηση. Καταρχάς πρέπει η ενημέρωση να δίδεται σε όλους δεν θα ζητήσει κανείς από μόνος του αυτή τη δυνατότητα. Η πρόσβαση, η ενημέρωση, η επικοινωνία με τον καταναλωτή είναι πάρα πολύ σημαντική για το συνολικό αντίκτυπο. Το δεύτερο πράγμα που έχει σχέση με τη σημερινή μας συζήτηση είναι ότι ε, οι επιχειρήσεις... Ε, οι λιανικοί πολιτές και ε, οι επιχειρήσεις πληροφορικής που τους υποστηρίζουν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ε, καταναλωτών. Διαφορετικά δεν μπορούν να υποβάλουν ε, τις σχετικές εκθέσεις. Πού είμαστε σήμερα στην Ευρώπη όταν υπάρχουν ε, αυτοί, αυτοί οι ενημερωμένοι λογαριασμοί, ε, η μείωση της κατανάλωσης είναι περίπου 3% κατά μέσο όρο. Αυτό που λέω είναι προσπαθούμε ε, να εισαγάγουμε τους ευφυείς μετρητές στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, οι περισσότεροι εκ των οποίων σήμερα δίνουν τη δυνατότητα μία ενημερωμένης τιμολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα θέματα που θα θέλαμε να καλύπτουν ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δαπανηρό να το επιτύχουμε με αυτούς τους μετρητές. Αν δηλαδή οι λιανοπολιτέ δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ε, των καταναλωτών δεν θα μπορούν να ε, δώσουν ε, όλα αυτά τα πράγματα στους καταναλωτές που θα μπορούσαν να δώσουν αν χρησιμοποιούσαμε πλήρως το δυναμικό των εφιών μετρητών. Αυτό βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, δηλαδή καταναλωτές Ενό τεραβάτ ηλεκτρισμού κατέτος ε, με τη μείωση που λέμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε υπάρχει μία μείωση 30 ε, μεγαβατόρων ε, μηνιαίως σε κάθε νοικοκυριό. Αν όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, γίνεται η εξοικονόμηση των 30 ΜΒ που σας είπα, ε, που σας ανέφερα. Διαφορετικά, μόνο 5% των καταναλωτών θα είναι αρκετά ενημερωμένοι για να ζητήσουν τέτοιου είδους προγράμματα. Ε, άρα οι πιθανότητές μας να επιτύχουμε το στόχο μας μειώνονται κατά 95%. Σύμφωνα με τις μελέτες των τελευταίων, των τελευταίων 7 ετών, βλέπουμε ότι η ενημέρωση, η πληροφόρηση είναι το πρώτο βασικό στοιχείο για να υπάρξουν προγράμματα ενεργειακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που θέλουμε να επιτύχουμε στην Ευρώπη. Ε, και μιλάω και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για ε, ξυπνότερη χρήση της ενέργειας και για όλους αυτούς τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να ενθαρρύνω την Επιτροπή σας να λάβουν αυτούς τους παράγοντες ε, υπόψη γιατί βλέπουμε τους τομείς ανησυχίας και, και προτάσεων, οι οποίες είναι εξιστοί, είναι καταρχάς ε, ε σαφής συγκατάθεση. οι καταναλωτές ε, στην Ιρλανδία για παράδειγμα σημαίνει ότι δεν θα έχουν αυτόματη πρόσβαση στους ε, στα δεδομένα τους, δηλαδή ότι θα έπρεπε να δώσουν σαφή συγκατάθεση στους ε, Ιανοπολιτές να δώσουν τα δεδομένα τους. Εμείς θα προτείναμε αυτή η σαφή συγκατάθεση να μην είναι τόσο στενή που να μπλοκάρει τα, τους καταναλωτές από τα ίδια τους τα δεδομένα, γιατί, γιατί τότε ε, πρέπει κάθε φορά να περάσει από μια επιχείρηση πληροφορικής ή από κάποιο λιανεοπολιτή. Η ανάγκη ορισμού των ανώνυμων δεδομένων και του αποκλεισμού τους από, τον, ε, από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε ε, να το κάνουμε αυτό, γιατί αν υπάρχουν ανώνυμα ναι, δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ε, ώστε να πείσουμε τους καταναλωτές πόση ε, ενεργειακή εξοικονόμηση μπορούν να κάνουν ε, αγοράζοντας, για παράδειγμα, ένα νέο καταψύκτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζέσικα. Τον λόγο έχει για 8 λεφτά ο Ασέντε, ο Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω κάποιες τα, τα πορίσματα του, project μας του Spion ε, είναι ένα ε, project μέδρα της Βρυξέλλες. Ε, χαίρομαι γιατί ακούσαμε την προηγούμενη ομιλία, διότι έτσι σας, αυτό το που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα σύστημα που θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο μεν, χωρίς να χρειάζεται όμως μια τράπεζα δεδομένων. Και αυτό είναι προς όφυλος ε, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Καταρχάς θα σας δείξω ότι υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις ε, ε, στην προστασία του, του απορρίτου. Ε, χρειαζόμαστε την προστασία του απορρίτου από τρεις προοπτικές. Δεύτερον, ε, ε, την privacy αυτή την θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να διαφυλαχθεί μέσω κάποιων κανόνων και όχι με την εφαρμογή της τεχνολογίας. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε δεν θα πρέπει να την λέμε privacy by design, αλλά privacy by policy και εν κατακλείδη οποιαδήποτε πρόταση για privacy by design εξαρτάται από τις αρχές ε, που διέπουν τον κανονισμό. Εάν οι αρχές ε, δεν είναι γερές αν θέλετε, δεν είναι ασφαλείς, ε, τότε δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την privacy by design. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε δηλαδή σε έναν αδύναμο κανονισμό. Επομένως, υπάρχουν όπως σας είπα τρεις προσεγγίσεις. Είναι συμμόρφωση, ε, ελαχιστοποίηση των δεδομένων ε, και προσδοκίες των χρηστών. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα, πώς θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι τέχνοκεντρικό, οργανοκεντρικό και εστιασμένο στον χρήστη. Δεν θα μιλήσουμε για νέους μετρητές και τα λοιπά και ρολόγια, αλλά όταν μιλάμε για έξυπνα δίκτυα, μην ξεχνάτε ότι τους υπολογιστές τους έχουμε εδώ και 60 χρόνια. Άρα δεν χρειάζεται να έχουμε συγκέντρωση των δεδομένων για να ε, προχωρήσουμε Χρειαζόμαστε καλό feedback, σωστό feedback για να ε, εξασφαλίσουμε, διασφαλίσουμε τους καταναλωτές, για να έχουμε αποδοτικά δίκτυα. Ε, θα πρέπει όλοι οι καταναλωτές ε, να... Μάλλον πιστεύουμε ότι ε, εάν συγκεντρώσουμε τα στοιχεία αυτές οι τράπεζες δεδομένων ε, ε, αρέσουν μόνο στους hackers, εάν υπάρχει κάποια διαρροή θα δημιουργηθούν προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Ε, υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες από τη στιγμή που εισήχθη ε, ο έξυπνος μετρητής στην Ευρώπη, το είδαμε αυτό και στην Ολλανδία. Ε, είχαμε προβλήματα, επομένως τα άτομα, οι πολίτες φοβούνται ότι κάποιος τους κατασκοπεύει, ή και μέσα στο, στην οικογένεια όλοι ξέρουν τι, ηλεκτρο, τι ηλεκτρικές συσκευές χρησιμεύει ο καθένας και πού και πότε κτλ. Επομένως, τι προτείνουμε σαν ερευνητές όσον αφορά το απόρριτο ή την προστασία του ιδιωτικού βίου. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι η... θέλουμε ε, να ε, θέσουμε τους πολίτες ενώπιον του διλήμματος ή θα έχουν ένα έξυπνο σύστημα ή δεν θα έχουν σύστημα καθόλου. Ε, εμείς θα θέλουμε να έχουμε μια καλή λειτουργικότητα χωρίς να έχουμε συγκέντρωση των δεδομένων. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ ε, είναι μια εταιρεία, 100 μέτρα ε, βλέπετε μετρητόνο, που, μιας προστασίας που προστατεύει τα, τα δεδομένα και κάνει αντίστοιχες έρευνες. Εδώ έχουμε όλα τα δεδομένα, τα μεμονωμένα δεδομένα, δεν συγκεντρώνονται όμως σε κάποια τράπεζα δεδομένων. Και έχουμε πληροφορίες για συγκεκριμένους σκοπούς. Επομένως, θα μας πείτε ποια είναι η λειτουργία την οποία θέλετε, θα συλλέγουμε τα δεδομένα, θα τα κρατάμε παράμερα και έχουμε την δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου. Προχωράμε επομένω. Θα ήθελα εν συντομία να σας μιλήσω για τα οικονομικά δεδομένα και ε, για την, ε, όσον αφορά τις διαφημίσεις που στηρίζονται στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Εδώ έχουμε κάποια κλικ που εμφανίζουν τις επιλογές ε, που έχει ο καταναλωτής ε, θα έπρεπε να, δω, να, σας προσφέ... να σας δω, δείξω ένα βίντεο, αλλά τέλος πάντων έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη διαφάνεια. Ε... έχουμε εδώ κάποιες, κάποιες, κάποιες επιχειρήσεις που ονομάζουμε trackers που λένε τι αυτοί ε, ανοιχνεύουν αν θέλετε, ποιες είναι οι συμπεριφορές και ποιες είναι οι αντιδράσεις σε κάποιες διαφημίσεις. Και μετά τα στοιχεία αυτά τα δίνουν σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις. μπαίνει ένα, κάποιο software στον υπολογιστή όπου μπορούν να ε, ανοιχνεύσουν την, ε, τις συμπεριφορές σας και την πόσο αντιμετωπίζετε τον υπολογιστή είναι σαν να υπάρχουν κοργοί τέλο πάντων στον, ε, στον υπολογιστή σας. Ε, τι συμβαίνει επομένως όταν ε, υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις, βλέπουμε ότι αυτές παρακολουθούνται, παρακολουθείται η αντίδραση και η συμπεριφορά του καταναλωτή. Τα κλίξη είναι πάρα πολύ σημαντικά και εφόσον μιλάμε για χρήματα, γίνεται μια, ε, υπάρχει ένα κίνητρο για ε, δόλια συμπεριφορά και για απάτες. Πολλοί ε, κάνουν κλικ και στις δικές τους διαφημίσεις για να κερδίσουν παραπάνω χρήματα και πολλές φορές πρέπει να πατήσετε κι εσείς οι ίδιοι σε κάποια διαφήμιση για να περάσετε στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Σε αυτή την απάτη του κλικ έχουμε και άλλη μία άλλη ε, απάτη. Προσπαθεί κάποιος να, κατα... να, να, να, να παρακολουθήσει κάποιον άλλον. Και έχουμε εταιρείε που κατασκοπεύουν όλους μας και εμάς και εσάς στο, στο ίντερνετ. Λοιπόν, δημιουργούμε με τον τρόπο αυτό διάφορες ε, τράπεζες δεδομένων που αναλύουν τη συμπεριφορά μας. Οι χρήστες ε, το καταλαβαίνουν αυτό και πολλές φορές ε, εξαφανίζουν τα cookies και πολλές φορές οι τράπεζες δεδομένων είναι απλώς μια συσσόρευση post data. Επομένως, αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι αν είχαμε σαφείς κανόνες ε, ε, προστασίας ε, των, του καταναλωτή και του, και του απόρριτου και των προσωπικών δεδομένων και μπορούσαμε να βρούμε αυτούς που παρακολουθούν τους καταναλωτές, πιστεύω ότι θα επηρεαζόταν η καθημερινή μας ζωή θα έπρεπε να συνοψίζω. Αυτή είναι η προσέγγιση της συμμόρφωσης που μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας και την τεχνολογία για να εξασφαλίσουμε ε, συλλογή πληροφοριών που είναι διαφανής και χρήσιμα και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Εδώ βλέπετε κάποιες, ε, κάποια λουλούδια τα οποία δείχνουν πόσο το προφίλ του Facebook είναι, γίνεται οικείο στους καταναλωτές ε, βλέπετε τι γίνονταν το 2005, ε, λίγες πληροφορίες, ε, το 2009 κάτι λιγότερες, ε, κάπως περισσότερες πληροφορίες ήταν πελάσιμες, Το 2010 σχεδόν όλες οι πληροφορίες είναι προσπελάσιμες. Βλέπουμε επομένω ότι υπάρχει και μία δυσαρέσκεια από πλευρά των καταναλωτών που συμμετέχουν σε αυτά τα websites. Επομένως υπάρχει και άλλη μια προσέγγιση που είναι η προσδοκία των χρηστών. Δηλαδή οι χρήστες πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα προστασία των δεδομένων που αντιμετωπίζουν ε, στο ίντερνετ. Τι πρέπει να κάνουν ε, αυτοί οι άνθρωποι για να προστατεύσουν ε, τα δεδομένα τους. Αλλά και θέματα κοινωνικού απορρίτου το προφίλ μου θα το δούνε οι, οι εργοδότες μου, οι γονείς μου, κάποιος, κάποιο άτομο το οποίο έχω δεσμό, μήπως αυτό παραβιάζει την ε, προστασία των δεδομένων. Ε, μπορεί να γελάτε, αλλά και ένας ε, μετρητής μπορεί να έχει στοιχεία για τα μέλη της οικογένειας και σε περίπτωση κάποιας φιλονικίας, κάποιας διαφοράς μπορεί να χρησιμεύσουν. Αυτές είναι τρεις προσεγγίσεις, η ελεγχιστοποίηση των και οι προσδοκίες των Χριστών. Ελπίζω να σας έπεισα ότι πρόκειται για ξεχωριστές προσεγγίσεις και πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι τρεις. Ε, μέχρι στιγμής η συμμόρφωση ήταν ε, η προσέγγιση η οποία εφαρμόζαμε περισσότερο για την προστασία των δεδομένων. Δηλαδή οι εταιρείε και οι επιχειρήσεις είχαν κάποιους κανόνες συμπεριφοράς, ε, σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις ήταν υπόλογες. Δεν γινόταν όμως καμία αλλαγή της τεχνολογίας και δεν ελαμβάνουν δεν ε, ε, ε, το υπόψη η προσδοκία του χρήστη. Ευχαριστώ. Τον λόγο τον έχει ο κύριος Κέλλη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Απλώς ήθελα να πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις ε, και μπορεί να παρουσιάζουν και στοιχεία που δεν θα ε, τα είχαμε σκεφτεί διαφορετικά. Ανάλογα με την πολιτική ιδεολογία του καθενός μπορεί να είναι διαφορετική και η προσέγγιση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας είναι να μην υπάρχει ένας φραγμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις ε, και ε, το όφελος των καταναλωτών σαν να ε, έπρεπε να αντιμάχονται το ένα το άλλο. Δεν σημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων πρέπει να βλάπτει τον καταναλωτή. Θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε. η εταιρεία που χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά και τα χρησιμοποιεί προ του καταναλωτή δεν πρέπει να μπαίνει ε, να παραβιάζει την προστασία των δεδομένων και να μπαίνει στον ιδιωτικό βίο του καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα κάπως να τα εξισορροπήσουμε. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ε, οι παρουσιάσεις αυτές είναι τόσο σημαντικά εργαλεία για μας, γιατί μας δίνουν πραγματική, ε, μια πραγματική οπτική γωνία και μας δείχνουν τι θα συνέβαινε εάν δεν λαμβάναμε υπόψη ε, τις ε, διάφορες ε, οπτικές γωνίες των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων που βλέπουν ακριβώς πώς η προτινόμενη νομοθεσία θα επηρέαζε τις επιχειρήσεις τους. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτά που μας είπατε και περιμένω εναγωνίως να δω τι θα πούν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντότερ έχει τον λόγο. Έχω μία ερώτηση για την Τζέσικα. η επιχείρησή σας, η εταιρεία σας προσπάθησε να ασχοληθεί με δεδομένα ε, συσσωρευμένα που δεν αφορούν τους καταναλωτές μεμονωμένα, διότι πολλές φορές ε, όσοι ασχολούνται με τους ε, ευφυείς μετρητές θεωρούν ότι είναι καλύτερα να ασχοληθούμε για, με γειτονιές και όχι με μεμονωμένους καταναλωτές. Ναι, είναι η σύντομη απάντηση. Ε, το ερευνήσαμε το θέμα. Εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος σας. Αλλά ένας ευφύης μετρητής θα μπορούσε να προσφέρει ε, στοιχεία ανά δευτερόλεπτο για την κατανάλωση κάποιου. Και αυτό ε, θα είναι σημαντικό για να, το, για να πάει στον ε, λιανοπολιτή τέλος πάντων. Αυτό όμως θα μπορούσε να είναι και παραβίαση των δεδομένων στις, στις αγορές ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, στον, του Καναδά, της Αυστραλίας ε, υπάρχουν στοιχεία οριέα τα οποία συσσωρεύονται και ξέρεις ένα αριθμό. Και το ξέρεις δηλαδή πρόκειται για ημερήσια κατανάλωση, για νυχτερινή κατανάλωση κτλ. δεν μπορεί να κάνει συγκρίσει ή να αντικαταστήσει την κατανάλωση του ενό με αυτή τον, του γειτονά του. Στην Γερμανία χρησιμοποιούν ε, την, ε, την κατανάλωση του γείτονα απλώς και μόνο για την ε, τιμολόγηση. Δηλαδή βλέπουν ότι ο ένας γείτονας πληρώνει πολλά, ο άλλος πληρώνει λιγότερα αλλά σαν feedback χρειάζεσαι στοιχεία για την δική σου κατανάλωση που πρέπει να γίνεται ε, σε, μηνιαία, σε ωριαία βάση. Ολοκληρώσαμε το πρώτο κομμάτι. Θα ήθελα να προσθέσετε κάτι. Ναι, να πω κάτι γρήγορα. Οι συνάδελφοι που έχουν απτύξει αυτή την τεχνολογία Μιλάμε για μεμονωμένα δεδομένα. Χρησιμοποιούν μια τεχνολογία, την κρυπτογραφία, που ε, τον, ε, στην επιχείρηση ότι έχεις ε, χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη ενέργεια, αυτήν και όχι ούτε παραπάνω ούτε λιγότερη. Τώρα, ε, συσσωρευμένα δεδομένα, ναι, όντω μπορούμε να δώσουμε συσσωρευμένα γεγονότα, α πούμε, για, τους, για τα ψυγεία. Αν μα το ζητήσετε, μπορούμε να το κάνουμε. Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είπε και η Τζέσικα είναι ότι δεν θα σας δώσουμε στοιχεία για σε καθημερινή χρήση. Θα σας δώσουμε ένα δείγμα, παραδείγματο χάρη, για κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Που, και νομίζω ότι αυτό σέβεται τις διατάξεις του κανονισμού. Γιατί σεβόμαστε και την προστασία των δεδομένων, αλλά και τις καλές εμπορικές πρακτικές. Να πω κάτι. Για τον καταναλωτή μπορεί να είναι συσσωρευμένα ή οτιδήποτε κρυπτολογία ή δεν, δεν, δεν τον ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Θέλουν να ξέρουν τι χρησιμοποιεί, τι χρησιμοποιεί ο ίδιος ο καταναλωτής. Απλώς εμείς θέλουμε τους ευφύς μετρητές να, ξέρει, να ξέρουν ε, οι καταναλωτές τι χρησιμοποιούν. Θα κοστίζει και 400 εκατομμύρια ευρώ το όλο project. Δισεκατομμύρια. Επομένως, ε, θα πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής τι χρησιμοποιεί. Συμφωνώ απόλυτα ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι προστατευμένα, δεν πρέπει να τα μπορεί να τα, να τα αγοράσει κάποιος, ε, θα πρέπει να είναι μεμονωμένα αλλά όχι υπερβολικά κατακαιρματισμένα. Ε, δηλαδή δεν πρέπει να προστατεύουμε τόσο πολύ τους ανθρώπους να μην ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν. Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα στο καταναλωτή, στον χρήστη. Απλώς δεν δίνονται, στον, στον κεντρικό σερβερ. Αυτό, αυτή δεν υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων που να υπάρχουν όλα τα στοιχεία να πάσα στιγμή. Αυτό είπα. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρο σου. Ευχαριστώ την Τζέσικα Στρόμπακα και την ε, κυρία Ντούρσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και τις δύο. Περνάμε στο επόμενο τμήμα, στο επόμενο κομμάτι της ε, ακρόασης. Δεν έχουμε πολλούς ε, συναδέλφους παρόντες, υπάρχουν ε, πολλές συνεδριάσεις φαίνεται. Ο πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριος Κρίστοφ Φίντλερ του European Magazine Media Association. Δέκα λεπτά έχει στη διάθεσή σας. Αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο κυρία Σαρτόρη και τον εισηγητή κύριο Κέλλη για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σα μιλήσω για μια πολύ σημαντική ανησυχία που έχει να κάνει το, με τον κανονισμό και την προστασία δεδομένων. Το direct marketing και ο ελεύθερο τύπο είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Για να καταλάβετε γιατί ανησυχούμε, θα πρέπει να σα δώσω μια ιδέα για τον τύπο σήμερα. Την κατάσταση. Βλέπετε εδώ κάποια περιοδικά, κάποιες εφημερίδες ε, και τις πλατφόρμες. Έχετε το μπλε που είναι έτυπος τύπος, ε, με το κίτρινο έχετε ε, σε διάφορα παιδιά Και στο τρίτο είναι τα σε Τι βλέπουμε λοιπόν από όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα κάτι πολύ θετικό, ότι υπάρχει μεγάλη επιτυχία εκδοτική στον τύπο, είναι ουδέτερη τεχνολογικά σήμερα, και, πληρώνει και μια, εκπληρώνει και μια δημοκρατική λειτουργία. Αλλά πιο ε, από το ίδιο το διάγραμμα υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να συναγάγουμε κάποια συμπέρασματα. Παραδείγματο χάρη το μπλε για τον τύπο. Βλέπουμε εδώ κάποια ε, στοιχεία που έχουν να κάνουν και με την χρηματοδότηση. Θα θέλαμε δηλαδή να υπάρξει ένα καλύτερο νομικό πλαίσιο για τον τύπο από του τη πολιτική ε, και επειδή δεν υπάρχει αυτό, προσπαθούμε να διατηρήσουμε το status quo. Από το διάγραμμα όμως καταλαβαίνετε ότι τελικά είναι όλο και πιο σημαντικό κάτι τέτοιο και αυτό ισχύει και για το άμεσο marketing. Τώρα, περιοδικά εφημερίδες χρειάζονται το άμεσο marketing και θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και η δημοσιογραφία. Θα σας εξηγήσω ε, το συνδρομητικό τύπο στη συνέχεια και για το συγκεκριμένο τον γενικό και τον ειδικό και την ε, κυκλοφορία. Δεν έχουμε βάλει τα τάμπλετ εδώ, βλέπετε μόνο τον έντυπο τύπο. Έως το 40% των συνδρομητικών περιοδικών και εφημερίδων εξαρτάται από την δυνατότητα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για στόχους άμεσου μάρκετινγκ. Πώς, λειτουργεί αυτό. Παραδείγματο χάρη στέλνει ένα περιοδικό για ποδήλατα, συγκεκριμένες ρυθμίσεις ε, ή μία συνδέση εφημερίδα στέλνει μέλη, ε, κάποια άλλα αλληλογραφία για μαγαζιά ρούχων για άντρες. Τα προσωπικά δεδομένα στέλνονται στον εκδότη που είναι ένας τρίτος και ο οποίος ε, επεξεργάζεται η τα φαντασία για τους ε, στόχους του άμεσου μάρκετ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να σταθμιστεί η διακύμαση, φυσική διακύμαση 30% των συνδρομητών ανά έτος, ανάλογα με τον τίτλο, ανάλογα με τον τομέα. Επομένως, οι εκδότες συνεχώς πρέπει να έρχονται σε επαφή με δυνητικά νέους αναγνώστες. Όχι τους ε, ήδη υπάρχοντες, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε αναγνώστες που δεν είναι ακόμη συνδρομητές και που θα ενδιαφέρονταν ίσως να γίνουν τακτικοί αναγνώστες, συνδρομητές, άρα χρειάζονται οι κατάλογοι διευθύνσεων από τρίτους για τους ε, εκδότες. Η συνδρομή λοιπόν πρέπει να εξηγηθεί ως ε, προϊόν. Χρειάζεται το άμεσο μάρκετινγκ, δεν υπάρχει πρατήριο πώληση. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να πω ότι υπάρχει μια παρανόηση ο νόμο περί δεδομένων ασχολείται μόνο με το πόσο και πού να χρησιμοποιηθούν κάποια δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση άμεσο μάρκετινγκ για συνδρομή σε περιοδικά εφημερίδε. Μπορεί τώρα να μπορεί για το άμεσο μάρκετινγκ να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία, οι διευθύνσει δηλαδή, αλλά υπάρχουν και κάποιε άλλε προποθέσει. Παραδείγματο χάρη για την τηλεφωνία, τηλεφωνικό μάρκετινγκ. Πολλέ φορέ χρειάζεται τον προτέρων συγκατάθεση. Για το email αντίστοιχα. Αλλά για να συνοψίσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τύπο ε, να έχει ε, επαφή ε, στα στοιχεία αυτά των συνδρομητών για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ. Αυτά τις λοιπόν πιστολές είναι σημαντικές και για τους παραλήπτες, όχι μόνο για τον τύπο και έτσι τα μειονεκτήματα αντισταθμίζονται θα έλεγα. Και αυτό το διαπιστώνουμε γιατί υπάρχουν πολύ λίγες ενστάσει. Οι περισσότερες είναι θετικές απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη, μία με δέκα είναι οι για 100.000 επιστολέ. Και να σα δώσω τώρα κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα εκδοτικό οίκο που αποκαλεί το Βέλγιο και τη Γαλλία, Group Express Roland, Ρτά με 800.000 συνδρομητέ. Κάθε χρόνο πρέπει να βρουν 310.000 νέους συνδρομητές και από τα direct mailings καταφέρνουν να έχουν το 42% αυτών των νέων. Και βλέπετε και κάποια άλλα στοιχεία για την Express ή για το Prospect. Στην πρώτη περίπτωση βλέπετε νέοι συνδρομητές 110.085 από τα direct mails και στο πρόσφυγε 25% και 60% προέρχεται από το άμεσο marketing. Στην Γερμανία, τις περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, το 20% περίπου της ε, κυκλοφορίας ε, των συνδρομητικών εξαρτάται από τα άμεσα από τις άμεσες ε, αλληλογραφίες, άμεσα mailings. Εδώ βλέπετε τώρα κάτι καινούριο, ίσως να μην είναι πολύ γνωστό. Αυτά τα ειδικά περιοδικά, ε, τα εξειδικευμένα, που έχουν ε, στόχο άτομα που απασχολούνται σε συγκεκριμένου ε, κλάδους και χρηματοδοτούνται ως καταναλωτικός τύπος είτε από συνδρομές, είτε από διαφημίσεις ή πώληση μέσω κάποιων περιπτέρων κτλ. Κυρίως και από τα δύο. Πρόκειται για ελεγχόμενη κυκλοφορία. Και η διανομή αυτή υπάρχει πάνω από 110 χρόνια ήδη. Δηλαδή, το 100% των ε, αντιτύπων αποστέλλονται σε εξειδικευμένους συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή βάσει συγκεκριμένων καταλόγων. Και θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα πεδίο, μια ομάδα στόχου, κάποιοι ειδικοί εμπειρογνώμονες και τότε θα μπουν και στο περιοδικό οι διαφημίσεις. η επεξεργασία των διευθύνσεων γίνεται με βάση το θεμητό συμφέρον. Υπάρχει το δικαίωμα ένστασης και οι επιχειρήσεις, οι οργανωτές κάποιων εκθέσεων τα κτλ. μπορούν να στείλουν τους καταλόγους στον εκδότη. Ενώ μια άλλη πηγή είναι κάποια μητρώα, το ίντερνετ κτλ. Αυτό ο εξακευμένο τύπο είναι πολύ σημαντικό στην το βασιστή στη γνώση, γιατί η ενημέρωση συνεισφέρει στην συνεχή επαγγελματική βελτίωση και εξέλιξη των αναγνωστών. Και πάλι εδώ βλέπουμε πολύ λίγες ε, ε, ενστάσεις. Εκατομμύρια θα έλεγα επαγγελματιών εκτιμούν τις πληροφορίε αυτές που λαμβάνουν. Εδώ θα σα δείξω κάποια παραδείγματα. Στι περισσότερε περιπτώσει είναι διαφορετικό ε, το μείγμα των συνδρομών και τη ελεγχόμενης κυκλοφορία, δηλαδή χρηματοδότηση μέσω διαφημίσεων. Το industry, πάλι από αυτό τον όμιλο Ρουλάρτα, βλέπετε 23 περίπου ε, αντίτυπα, βλέπετε πολύ λίγες συνδρομές. Στο Data News όμως βλέπουμε περισσότερες συνδρομές, σε 15% και 85% ελεγχόμενη κυκλοφορία και για τη Γερμανία βλέπουμε το Car Industry περίπου 90% ελεγχόμενη και 10%, 11% συνδρομή. Το Process Industry και άλλα παραδείγματα. Machine Market, 89 ελεγχόμενοι, 11 συνδρομή. Ένα άλλο για τρόφιμα, βλέπετε τα στοιχεία, 36 περίπου ελεγχόμενοι, 6% συνδρομή. Και τελευταίο, το περιοδικό Painter που εδώ βλέπουμε 22% συνδρομή, 74% ελεγχόμενη κυκλοφορία. Άρα, ο τύπος, ε, όλοι οι κατηγορίες ε, ουσιαστικά είναι να έχουν ως μέλημα να διατηρηθεί η προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το άμεσο μάρκετινγκ και ιδίως για τον εξειδικευμένο τύπο, αλλά και για τις εφημερίδε και τα περιοδικά και περιλαμβάνει και τη διαθεσιμότητα καταλόγων διευθύνσεων από διάφορε πηγέ. Άρα οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να δίνουν τι διευθύνσει στου εκδότε αλλά με βάση το θεμητό το νόμο συμφέρον του τρίτου μέρους, του εκδότη. Και θα πρέπει να είναι αναλογικές οι προϋποθέσεις για την ε, παροχή των πληροφοριών και να μην ε, συνιστούν ε, άχθος. Γιατί αν πια είναι πάρα πολύ αναλυτικό, πολλέ λεπτομέρειε δεν είναι πλέον και αποδοτικό. Ψηφιακά λοιπόν επιχειρηματικά μοντέλα και αυτά δεν θα τα αναλύσω. Θα πρέπει να σας πενθυμίσω όμως απλά ότι θα πρέπει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τις έχουμε υπόψη μας. Δεν θα πρέπει να βρεθούν σε μειονέκτημα απέναντι σε μεγάλες επιχειρήσεις που κυρίως ε, στα επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται. Έχουμε το lock-in και το opt-in, αλλά όταν πάμε στην, στα σελίδα μιας ε, μικρής, ε, ε, ένας μικρός εκδοτικού οίκου θέλει κανείς να διαβάσει μόνο το άρθρο. Πάντως, όπως και να έχει. Χρειαζόμαστε τις ευκαιρίες, χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τη ε, δημοσιογραφία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Νομίζω τώρα μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο μιλητή τον κύριο Τζόζεφ Αλάντεφ από την Oracle. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Κέλλη και τους οργανωτές της σημερινής ακρόασης. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να υπενθυμίσω πηγαίνοντας μερικά χρόνια πίσω σε έναν από τους λόγους για τους οποίους ασχοληθήκαμε με την ανάγκη μιας νέας οδηγίας και ήταν η αλλαγή περιβάλλοντος ε, που υπάρχει γύρω μας, το πλαίσιο δηλαδή, στο πλαίσιο, στο, πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η οδηγία το cloud computing, ε, το ίντερνετ, ε, η ψηφιακή οικονομία και η εξάπλωση των υπηρεσιών μεταξύ διαφόρων χωρών, ε, μεταξύ διαφόρων δικτύων διανομής γίνονται πλέον οι υπηρεσίες. Άρα οι καταναλωτές έχουν πολύ περισσότερους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα. Υπάρχει, μεγαλύτερη, υπάρχει μια μεγαλύτερη ροή ε, νόμων προστασίας του ιδιωτικού βίου, όπως επίσης και η ανάγκη ύπαρξης οικονομικής ανάπτυξης, ε, απασχόλησης ε, και ασφάλειας δικαίου. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι ο βασικός στόχος πίσω από το σχέδιο κανονισμού ε, ήταν ε, κοινή και θετική, δηλαδή πιο αποτελεσματική νομοθεσία, με την οποία συμφωνούν οι εμπλεκόμενοι ε, ε, φορείς, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη εναρμόνιση, χαμηλότερο ε, διοικητικό άχθο, εξοικονόμηση κόστους, επισήμανση των υποχρεώσεων επειδή γίνεται πιο περίπλοκος πλέον ο κόστος μας, να είμαστε βέβαιοι επίσης ότι μπορούμε να έχουμε πολλαπλέ λύσεις οι οποίες όμως είναι ευέλικτες και επίσης ε, οι κώδικες δεοντολογίας είναι πολύ σημαντικοί σε αυτό το πλαίσιο, το πλαίσιο ε, και επίσης μελέτες αξιολόγησης αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων σε ε, πολλές περιπτώσεις δηλαδή οι στόχοι της νομοθεσίας ήταν κοινοί για όλους και νομίζω ότι σε, μέρη, σε γενικές γραμμές θεωρήθηκε ότι καλά ήταν όλα αυτά όμως είναι πολύ δύσκολο να τα επιτύχουμε και το να υπάρξει ε, μία νομοθεσία στην οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι πραγματικά μία μεγάλη πρόκληση. Όταν βλέπουμε λοιπόν μερικέ, μερικά από τα σημαντικά ωφέλη και θα ήθελα να πω ότι όταν μιλάμε για κάποιες αδυναμίες που μπορούν να υπάρχουν στο σχέδιο νομοθεσίας, στο σχέδιο κανονισμού, θα αναφερθούμε και σε, ορισμένες, ε, σε ορισμένα στοιχεία τα οποία το Κοινοβούλιο ήδη κάλυψε. Παρ' όλα αυτά θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ε, τα ε, ε, θέσουμε χωρίς να πούμε πώς τα αντιμετώπισε η κάθε επιτροπή. Όταν θέλουμε λοιπόν να μεγιστοποιήσουμε το όφελος από απόψεως επιχειρηματικής, το μεγαλύτερο μέγεθο, όφελος είναι αυτό το one-stop shop ή τέλο πάντων η βασική αρχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο επιχειρήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση ώστε αυτό να είναι σαφές. Όμως ε, είναι γεγονός ότι η προσπάθεια ε, γίνεται και ε, ως τέτοια εκτιμάται. Επίσης έχει σημασία πού βρίσκεται η κάθε επιχείρηση, γιατί κάποια πολυεθνική μπορεί να έχει ένα κεντρικό γραφείο, να έχει κεντρικά γραφεία σε, σε πολλές χώρες, οπότε ο ρόλος της χώρας στην, ύπαρξη, στην αναγνώριση της βασικής εγκατάστασης επιχείρησης είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η κύρια αρχή και πρέπει επίσης να μπορούμε να πάμε στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων όταν υπάρχει κάποια παραβίαση, να ξέρουμε δηλαδή σε ποιον θα απευθυνθούμε, όμως πρέπει να υπάρχει μια, ένα συντονισμός και μια συνεργασία προκειμένου να λυθούν ε, οι διαφορές. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ε, οι εταιρικοί κανόνες ε, αναφέρονται σαφώς ε, μεταφορές ε, ε, η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των, των βασικών αρχών των διαφόρων επιχειρήσεων πρέπει να διευκολυνθεί. Μπορεί να υπάρχουν ίδιες παρόμοιες λύσεις, εν πάση περιπτώσει, για παρόμοιου τύπου επιχειρήσεις. Επίσης υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στο πώς ε, θα, υπα... θα αποσαφινιστεί ο ρόλος του ελεγκτή και του επεξεργαστή. Δύσκολα είναι εδώ τα πράγματα γιατί είναι διαφορετικές οι αξιώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαφορετικές ε, αυτές των Ευρωβουλευτών και πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα επιβολής των σημαντικών ε, απαιτήσεων των ελεγκτών και των επεξεργαστών, όμως δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τη σχέση αυτών των δύο. Επίσης, όταν αρχίσουν να υπάρχουν ε, ανεξάρτητες υποχρεώσεις ε, για τον επεξεργαστή, τότε ο επεξεργαστής πρέπει να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις πληροφορίες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ερχόμαστε πάλι στο θέμα της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του ρόλου του ελεγκτή, κάτι το οποίο δεν θέλουμε υποχρεωτικά να κάνουμε. Και επίσης το θέμα της, ε, της κοινής και εξ ολοκλήρου ευθύνη, κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τον επεξεργαστή και δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει μια τέτοιου είδους λύση. Τώρα, εξοικονόμηση κόστους και διοικητικό άχθος και αυτά ε, είναι στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να βελτιωθούν στο σχέδιο του κανονισμού, ε, διαγραφή ορισμένων ε, απαιτήσεων κοινοποίηση, θα μείωνε όντως το διοικητικό άχθος και το, την εξοικονόμηση του κόστους, όμως δεν γίνεται αυτό στο βαθμό που βλέπουμε στην οικονομική ανάλυση. Μερικές φορές πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και αύξηση κόστους. Για, γιατί το λέω αυτό, γιατί μέχρι να ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή αρχίσει να λειτουργεί ο κανονισμός, δεν θα μπορούμε να ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η κατάσταση. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του επίπεδου της τεκμηρίωσης ε, που ε, πραγματεύονται πολλές ε, ρήτρες. Πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικές οι αναφορές σε αυτό το θέμα. Οι λεπτομέρειες δηλαδή που ε, ζητούνται είναι υπερβολικές. Η προηγούμενη διαβούλευση και έγκριση, η πρώτερη έγκριση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω ε, κόστος ε, και δεν ξέρω μάλιστα εάν είναι ανάλογη αυτή η αύξηση του κόστους με το όφελος που προκύπτει για την προστασία του δεδομένου. Όσον αφορά τώρα τις 24 ώρες για την κοινοποίηση της παραβίασης. Υπάρχουν όμως ορισμένες δραστηριότητες που είναι εκτός του ελέγχου του ελεγκτή. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα καθαρά πρακτικά ως προς αυτό. Ένα ακόμη θέμα είναι η επιχειρησιακή δυνατότητα, πώς δουλεύουν δηλαδή τα πράγματα. Έχουμε μιλήσει για το ρόλο της ε, αξιολόγησης αντικτύπου Ξέρουμε ότι αυτό προέκυψε από τη διαδικασία RFID ε, αρχικά ήταν ένα εσωτερικό έγγραφο, δεν ήταν ένα έγγραφο που αφορούσε την συμμόρφωση και με το να αφορά τη συμμόρφωση ε, ουσιαστικά αντιστρέφουμε τα πράγματα και δεν, ε, δεν επιτυγχάνουμε το στόχο που θέλουμε. Γιατί αυτό αρχικά, επαναλαμβάνω, ήταν ένα εσωτερικό έγγραφο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι πολύ σημαντικά αυτά τα έγγραφα ε, και ότι δεν πρέπει να είναι προσπελάσιμα από τον ελεγκτή, όμως πρέπει να γίνεται για επιτόπου, σε περιπτώσει επιτόπου ελέγχου, έρευνας ή αξιολόγησης ε, της ε, συμμόρφωσης. Όταν επίσης βλέπουμε το θέμα του privacy by design και της ασφάλειας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Είναι δύσκολο να τα επιβάλλουμε τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια, μια δομή στο πλαίσιο μιας οργάνωσης. Τώρα όσον αφορά την ασφάλεια υπάρχουν παγκόσμια πρότυπα ε, που χρησιμοποιούν ε, μεγάλες, ε, μεγάλοι οργανισμοί και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνώμονας. Όμως Νομίζω ότι το ε, νομίζω ότι ο κανονισμός δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ λεπτομερής ε, ως προς την ε, ευελιξία της εφαρμογής. Θέλουμε να δούμε, πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στην εταιρεία να αποφασίσει εκείνη πώς θα τα εφαρμόσει και όχι να τις πούμε τι ακριβώς θα, πώς ακριβώς θα προβεί στην εφαρμογή. Ακούσαμε από τα FEE e δίκτυα κάποιες προβλέψεις για τον αντίκτυπο της νομοθεσίας αυτής. Πρέπει να αυξήσουμε τον αντίκτυπο ε, στον τομέα ε, της ιατρικής φροντίδας, της περίθελψης, ε, της ευφυούς χρήσης ενέργειας. Ναι, σε αυτούς τους τομείς όντως θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση λόγω του κανονισμού και πρέπει να δούμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε το όφελος αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε, μπορούμε να έχουμε και ε, όφελος για τους καταναλωτές και προστασία των δεδομένων. Το θέμα είναι πώς θα μεγιστοποιηθούν και τα δύο χωρίς να αντιμετωπίζουν, να αποτελούν το ένα πρόβλημα για το άλλο. Πρέπει ένα καθεστώς ε, να είναι αξιόπιστο, να είναι βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που ισχύει τώρα. Και επίσης πρέπει να δούμε ε, πώς από αποτρεπτικά ορισμένα πράγματα κατέληξαν να αποτελούν, να είναι στρεβλά ε, ίσως λόγω του πώς ακριβώς ε, είχαν πλαισιωθεί τα πράγματα. Επίσης χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ευελιξία στην εφαρμογή και θα ήθελα να ολοκληρώσω με δύο στοιχεία. Πρώτον, πρέπει να προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε τον κανονισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται καθαρά οι στόχοι πρέπει οι επιχειρήσει να συμφορφώνονται με τον νόμο, αλλά ο νόμος δεν θα έπρεπε να επιβάλλει υποχρεώσεις που είναι άχρηστες και πάρα πολύ λεπτομέρειε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βρεθεί αυτή η ισορροπία την οποία μίλησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρεμβάσεις. Ο συνάδελφος Κέλφιν να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ και στον Κρίστοφ και στον Τζόζεφ για αυτή την τόσο καλή και συνεκτική παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για μας. Απλώς να ρωτήσω μια-δυο ερωτήσεις. Πρέπει να προσεγγίσουμε νέους αναγνώστες και τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν που αποδεικνύουν ότι θα πρέπει να ε, βρίσκονται νέοι αναγνώστες για να διατηρεί το κλάδο σου. Και προσπαθούν να διατηρήσουν το status quo, από ό,τι κατάλαβα αυτή τη στιγμή. Οι προτάσεις ε, ε, πώς θα εξελιχθούν, διότι όταν βρίσκουμε κάτι καινούριο μετά από 10-15 χρόνια, πρέπει να ενδυναμώνουμε το status quo. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μία δράση έτσι ώστε να ενισχυθεί η όλη διαδικασία. Επομένως, μήπως θα μπορούσε ο συνάδελφος να μπει λίγο, λίγο περισσότερα. Ο Κρίστοφ, από τον Κρίστοφ ε, περιμένω. Επίσης, ο Τζόζεφ μίλησε για την μελέτη αντικτύπου που έχουμε στο Κοινοβούλιο για την Ήτρε που θα υποβληθεί, θα παρουσιαστεί αύριο υπό το φως των προτάσεων της Κομισιόν. Δεν μπήκε όμως σε πολλές λεπτομέρειες για κανένα από τα σημεία τα οποία έθιξε όσον αφορά τις συνέπειες στον αντίκτυπο. Επομένως, ήθελα να ρωτήσω για το διοικητικό κόστος και για τις οικονομίες. Πιστεύει ότι οι γενικές γραμμές, οι προτάσεις έτσι όπως έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής θα είναι αντιπαραγωγικές και θα, τελικά θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Για την, όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, στην εξοικονόμηση χρημάτων, περιορισμό του κόστους και να, και ε, να εμποδίσουμε την ανάπτυξη νέων μορφών τεχνολογίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η νομοθεσία έτσι όπως προτείνεται τώρα θα αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην Ευρώπη και όχι να τις ε, ενθαρρύνει όπως θα είναι ο σκοπός. Γιατί εάν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις στην ε, Ευρώπη, τότε θα περιοριστεί και η ανταγωνιστικότητά μας. Αν κατάλαβα καλά, ε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε με λίγα λόγια τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ ο, η συνάδελφος Άντρ Η πρώτη ερώτησή μου αφορά τους εκδότες οι κανόνες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι περίπου σαν και αυτούς τους που ισχύουν στη Γερμανία. Η εκδοτική βιομηχανία όμως στην ε, Γερμανία είναι ανθυρή. Επομένω, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί οι κανόνες ε, που θα επιβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι επιβλαβείς, ενώ στη Γερμανία ήδη οι κανόνες είναι, είναι καλοί. Τώρα, ερώτηση προς τον κύριο Άλαντεφ. Μήπως ε, θα έπρεπε να έχουμε ε, την ίδια αρχή προστασίας των δεδομένων ε, που έχουμε σε εθνικό επίπεδο και εδώ. Γιατί με τον τρόπο αυτό άρεται η, η αμφιβολία για το ποια αρχή προστασίας των δεδομένων θα αναλάβει δράση σε κάθε περίπτωση ο κύριος Φίντλερ. Να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση. Όπως σας προσπάθησα να εξηγήσω στη Γερμανία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη, ο τύπος είναι παρόν και είναι επιτυχημένος όσον αφορά την ε, ε, προσπελάσιμότητά του στους αναγνώστες. Βέβαια, παράλληλα υπήρχαν πολλές εφημερίδες που έπρεπε να κλείσουν τον τελευταίο καιρό. Και ο προτινόμενος κατοσμό προστασίας των δεδομένων θα είναι παρόμοιος με αυτόν της ε, γερμανικής που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία. Όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο είναι διαφορετική η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι ισχύει στην Γερμανία για την προστασία των δεδομένων και για την ε, ε, ε, μεταφορά δεδομένων, αν θέλετε, για την επαφή του B2B ή και η προστασία στον χώρο εργασίας επίσης. Εμείς κάναμε κάποιες προτάσεις και το πιο σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με την ισχύουσα γερμανική νομοθεσία που δεν λέω ότι ο πλευρά εκδοτών είναι η καλύτερη νομοθεσία του κόσμου, είναι μία από τις εκδοχές με τις οποίες μπορεί κανείς να ζήσει, αλλά η τελευταία μεταρρύθμιση που έγινε είναι τόσο περιορισμένη που εάν με ρωτούσατε ιδιωτικά και όχι εδώ, δημόσια, θα σας έλεγα ότι πολλά από αυτά τα οποία θα έπρεπε να γίνουν δεν μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τη γερμανική, γερμανική νομοθεσία. Ένα πράγμα όμως είναι σαφές ότι τα, τρίτο, τρίτα μέρη οι μπορεί, μπορούν οι βιβλιοπόλεις ας πούμε να κοινοποιήσουν τους καταλόγους των πελατών στους εκδότες και αυτό δεν φαίνεται τόσο σαφώς στο σχέδιο κανονισμού, διότι το συμφέρον του τρίτου μέρους δεν εμφανίζεται με τόσο σαφή τρόπο όπως στην οδηγία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που αφορούν την ε, υποχρέωση ενημέρωσης και μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αν θέλετε μετά την συνάντηση ή μέσα στα πλαίσια μιας άλλης συνάντησης μπορούμε να, συζητήσουμε, να συζητήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Επομένως το status quo, όταν μιλάω για status quo, μιλάω για τους εκδότες που έχουν ένα διαφορετικό, μια διαφορετική δομή στην Ευρώπη, αλλά μπορεί κάτω από συνθήκες συγκεκριμένες ε, τα τρίτα μέρη να μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους εκδότες για να αγγίξουν νέους ε, αναγνώστες ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα και επαναλαμβάνομαι εδώ είναι ότι θα πρέπει να διατηρούμε το συμφέρον του τρίτου μέρους και μετά θα πρέπει να δούμε ε, δεδομένα που αφορούν το προφίλ ε, ε, όταν πρέπει να δώσεις πληροφορίες δίνεις τις πιο σημαντικές πληροφορίες εφόσον υπάρχει αρκετός χρόνος ας πούμε ή Ίσως ε, πρόκειται για δεδομένα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Θα πρέπει επομένως να, να είμαστε σίγουροι ότι το direct marketing επιτρέπεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο όταν σκεφτείτε τις εξαιρέσεις από το direct marketing για τον τύπο. Είχαμε στην Γερμανία μια συζήτηση μέσα στα πλαίσια της τελευταίας μεταρρύθμισης και δεν το κάναμε αυτό, διότι η αγορά θα συρρυκνώνεται τόσο πολύ που θα χάναμε την δυνατότητα να ε, ε, αγγίξουμε, αν θέλετε, αυτούς τους, ε, τους ενδιαφερομένους κατά από κανονικές συνθήκες. Ευχαριστώ, κύριε Τζόζεφ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορώ να προσπαθήσω να απαντήσω και τις δύο ερωτήσεις από εκείνου γιατί σχετίζονται με τον τύπο. Αν δούμε, παραδείγματος χάρη το δεύτερο ερώτημα που λέει ότι βασική αρχή πρέπει να είναι και όπου έρχεται τα δεδομένα, η απάντηση είναι όχι. Τι μιλάμε εδώ. Μιλάμε για την βασική αρχή, για την ε, επιχείρηση που εξοικειώνεται σιγά σιγά με τις ε, πρακτικέ του Επιτρόπου σας των δεδομένων. Ο επίτροπο αυτό σιγά σιγά εξοικειώνεται και με την επιχείρηση. Επομένω, υπάρχουν καταγγελίες, αλλά ήδη έχει διαμορφώσει κάποιο υπόβαθρο. Ο Επιτρόπος και υπάρχει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη σχέση των δύο και λιγότερη ε, αλληλεπικαλυπτόμενη προσπάθεια όταν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός είναι κανονισμός δεν μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο. Ισχύει ανά την Ευρώπη το ίδιο αυτό ο Επίση, ο κανονισμό έχει και ένα μηχανισμό συνεκτικότητα. Άρα και η... το λεγόμενο forum shopping έχει περιοριστεί πάρα πολύ σημαντικά στην νομοθεσία. Δεν προτείνουμε βέβαια αποκείμενος αυτός να πηγαίνει στον Επίτροπο Προστασία Δεδομένων, ο οποίος δεν θα έχει λόγο για την επίλυση της διαφοράς. Θα έχει ρόλο, αλλά θα συνεργάζεται με την βασική αρχή και μαζί θα λύνουν το πρόβλημα. Έτσι, είμαστε δίκαιοι προς όλους και προς το υποκείμενο και προς ε, την, <coughs> Συγγνώμη, και προς την επιχείρηση. Άρα ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση, να έχουμε κερδισμένους μόνο. Ευρύτερα τώρα. Αν βγάλουμε και προσθέσουμε, τέλος πάντων, πού φτάνουμε, ποιο είναι το σύνολο. Εξαρτάται, αυτή είναι η απάντηση, εξαρτάται από την ε, νομοθεσία που θα δημιουργήσουμε. Γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και συνθήκες ε, που θα κάνουν μικρότερο το όφελος από το κόστος. Πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι το επίπεδο υποχρέωσης, το επίπεδο λεπτομέρειας που είναι γενές σε αυτά τα έγγραφα. Εκ των προτέρων έγκριση συγκατάθεση κτλ. Αυτοί οι παράγοντες ε, θα έχουν και πρωτογενή και δευτερογενή επίδραση. Και αν δεν υπάρχει έλεγχος, τότε δεν θα υπάρχει όφελος στη διαπραγμάτευση. Άρα, ουσιαστικά το θέμα είναι και η γλώσσα και η εφαρμογή και η ερμηνεία, ώστε να υπάρχει ευελιξία για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τις διαδικασίες τους. Και έτσι θα υπάρχει και η απαραίτητη αξιοπιστία και για τους καταναλωτές, δηλαδή να πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματική νομοθεσία η Ευρώπη επίσης πρέπει να είναι ανταγωνιστική και σε ό,τι αφορά την προσαρμογή σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες τεχνολογίες. Να αποκομίσει ωφέλη δηλαδή από όλα αυτά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση κάπως ε, παλαιομοδίτικων μορφών ε, άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κτλ. Βέβαια δεν σημαίνει ότι τα πετάμε αυτά και δεν μας ε, επηρεάζει καθόλου ούτε μας απασχολεί ο έλεγχος του ιδιωτικού βίου, αλλά το θέμα είναι ποιε είναι όλες το σύνολο των συνθήκων εντό των οποίων ε, θεσπίζουμε αυτούς τους ελέγχους. Μπορούμε να δούμε και κάποιε πτυχέ του σχεδιασμού, του design. Και πρέπει να είναι θετικές αυτές οι πτυχέ. Μπορεί το, το privacy by design να το βελτιώσουμε, χωρίς να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο βάρος. Αν έχουμε ένα πρότυπο κοινό όμως, template, τότε μπορεί να δημιουργηθεί βάρος επιπρόσθετο. Στόχος είναι να επικεντρωθούμε όχι τόσο στο πώς, αλλά στο τι. Για να μην δημιουργήσουμε περιορισμούς. Είναι λάθος να νομίζει κανείς ότι μία είναι η λύση, μία είναι η προσέγγιση και αυτό βέβαια έχει να κάνει και τελικά με αύξηση του κόστους. Grazie, bene, se non c'è... Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχει κανείς άλλος που ζητάει το λόγο, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Ευχαριστούμε... Α, α ο κύριος Κέλλη θέλει να προσθέσει κάτι ή θέλει να ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις διευκρινήσεις που έδωσαν. Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Οι ομιλητέ, κάποιος από τους ομιλητέ θεωρεί ότι ο πρωτονόμινος κανονισμός πλήττει ή εμποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων B2B σε σχέση με το B2C και Τζόζεφ για το πώς και όχι το γιατί. Εδώ ζητάς εσύ να υπάρχει μία περαιτέρω βεληξία στον κανονισμό που θα επιτρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα αυτού, αυτής της φύσης και θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν γίνει αυτό για την ανάπτυξη και για τους ε, καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Θα απαντήσω και τα δύο. Και στα δύο. Συμφωνώ απόλυτα με την διατύπωση που είπατε για το πώς και το τι. Εάν εστιάσουμε στο τι και υπάρχει ο κανονισμός, το πώς θα αντιμετωπιστεί μόνο του. Υπάρχει τεχνολογία η οποία θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο ευέλικτοι στο μέλλον. Τώρα, για την άλλη ερώτηση, σε B2B επίπεδο είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι από το B2C και δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τον κανονισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο πιο μεγάλο είναι το επίπεδο διαφοροποίησης, τότε θα είμαστε σίγουροι ότι οι υποχρεώσεις ε, ταιριάζουν με τις απαιτήσει και όχι ένα μοντέλο το οποίο να ταιριάζει σε όλους, διότι εκεί θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. αν δεν υπάρξουν περαιτέρω τροποποίηση στον κανονισμό, νομίζουμε ότι θα μπορούσε πραγματικά να βάλει σε κίνδυνο σημαντικά επιχειρηματικά μοντέλα για το B2B και το B2C. Είπαμε ότι είναι ουδέτερο τεχνολογικά ο τύπος. λάσων, γι' αυτόν θα έχει κάποια, κάποιο αντίκτυπο. When I'm, when I'm looking... Βλέποντα τα άρθρα εδώ, βλέπω ότι υπάρχουν πράγματι τομείς όπου, για παράδειγμα, τα ανωνυμοποιημένα ε, δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δουν επιχειρήσει να χρησιμοποιούνται λιγότερο ή περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και υπάρχουν και τα θεμητά συμφέροντα κτλ. Αν αυτά τα έχουμε περιορίσει, τότε κλείνουμε την ε, αγορά ουσιαστικά. Όπως πολύ σωστά είπε ο Τζόζεφ, δεν είναι απλό ότι υπάρχουν, είναι πώς ορίζονται, πώς διατυπώνονται. Okay, well, um, I think... Τρεις προσεγγίσεις, ε, ελαχιστοποίηση, συμμόρφωση και τα λοιπά, τα τρία αυτά που τις προσεγγίσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια ενοποίηση. Αν θέλουμε να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων B2B, μπορεί να χρησιμοποιείται προσέγγιση της συμμόρφωσης και ο Τζο έχει πολυετή εμπειρία για αυτό το τομέα. Και για τη συμμόρφωση και για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων. Πώ όμω θα υπάρχει διαφάνεια προ τον καταναλωτή, ώστε να συμμετέχει ουσιαστικά στη διαδικασία, να μην ε, είναι μέσα σε αυτό το χάο που βλέπει και νιώθει χαμένο αυτή τη στιγμή. Πολλές λοιπόν μελέτες ε, χρηστών λένε συνήθως ότι δεν τους ενδιαφέρει τους χρήστες ε, η προστασία των ιδιωτικών δεδομένων το έχουν καταλήψει, γιατί είναι θέμα πιο πολύ τη αξιοπιστία, τη εμπιστοσύνη, τη δέσμευση σε κάποιε επιχειρήσει, σε κάποιε οργανώσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προσέγγιση, privacy by design, είναι σημαντική. Να βλέπει ο καταναλωτή τι γίνεται και με το B2B. Έχει έλεγχο. Πώ ρέουν τα δεδομένα μεταξύ των φορέων. Μήπως τον βαρύνει υπερβολικά η ευθύνη τελικά, να υπάρχει μια εξισορρόπηση ανωνυμοποιημένα δεδομένα. Ίσως μια κεντρική δήλωση είναι ότι εμείς ε, έχουμε δει πολύ αδύναμες σειρέ δεδομένων ε, ανωνυμοποιημένων. Δηλαδή μπορούν να εντοπιστούν, μπορεί να εντοπιστεί ταυτότητα, να γνωριστούν αυτά τα άτομα, να βγουν τα στοιχεία τους ε, και δεν μπορούν να έχουν προστασία. Επίσης μπορεί να υπάρχει παραβίαση, ακόμη και αν είναι ανωνυμοποιημένα τα δεδομένα. Εμείς αυτό που θα θέλαμε λοιπόν θα ήταν να υπάρξει κατανόηση της τεχνικής αυτής ε, εξέλιξης με την ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν είναι ανωνυμοποιημένα μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει, γιατί βλέπουμε κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις τελικά να μπορούν να έρθουν στο ύψος της πρόκλησης με την ανωνυμοποίηση. Μπορεί να γίνει αυτό λοιπόν. Έχουμε την ευκαιρία, δεν το έχουμε δει. Ελπίζουμε λοιπόν να ληφθεί σοβαρά υπόψη προσέγγιση αυτή. Ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η, η απογευματινή αυτή συζήτηση. Ήταν διαφορετική, υπάρχει, υπήρξε μεγαλύτερη ευελικτία, πιο ελευθερία στις παρεμβάσεις. Μην νομίζετε ότι αυτό θα επαναληφθεί και στο μέλλον. Αυτό έγινε και παραβιάσαμε τους κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής, διότι δεν είχαμε πολλούς συναδέλφους παρόντες και αποφεληθήκαμε από αυτή την κατάσταση. Έδρα επενθυμίσεις να στους συναδέλφους ότι αύριο ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, ότι στις 23 και 24 Ιανουαρίου θα έχουμε την συζήτηση για, την, για τις τροπολογίες και με βάση το χρονοδιάγραμμά μας θα περάσει από την Επιτροπή μας στις 21 Φεβρουαρίου. Θα περιμένουμε 5 λεπτά για να έρθει η συνάδελφος, ε, κύριος συνάδελφος ε, Σούζα Βάγνερ, που ήταν ε, παρόν προηγουμένως αλλά έπρεπε να φύγει. Λοιπόν, πέντε λεπτά ε, διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε στις 5 και τέταρτο λέει η πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να υπενθυμίσω στις παρούσες πολιτικές ομάδες να ενημερώσουν, να ενημερώσουν τους συντονιστές ότι μάλλον θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και πριν τις 6, αν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, ε, διάταξης, όπου η συγητής ε, είναι ο συνάδελφος Σόζα Βάγνερ και αφορά την τροποποίηση οδηγία 2003-87 με στόχο την διευκρίνηση των διατάξεων που αφορούν το χρονοδιάγραμμα των πληστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο συνάδελφος Σόζα Βάγνερ. Χωρίς μικρόφωνο, συνάδελφο. Σόζα Βάγνερ. Περδόν. Ε, συγγνώμη. όπω είπε η Πρόεδρο, είμαστε εδώ να συζητήσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το χνοδιάγραμμα των πληστηριασμών των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. Είχαμε κάνει πριν από κάποιες τη επιτροπή μα μια πρώτη προσέγγιση και είχα πει τότε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι εύκολα μπορεί να επιληθούν. Το πρώτο πρόβλημα είναι η αρμοδιότητα της Επιτροπής για να ρυθμίζει ε, αυτό το τομέα αλλάζοντας την υφιστάμενη οδηγία. Ε, νομίζω ότι είναι προφανές ότι η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα και αν μπούμε στον κόπο και διαβάσουμε και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Οικαστηρίου του Λουξεμβούργου, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα εκπομπών, που είναι άφθονη και ενδιαφέρουσα, βλέπουμε ότι οι δικαστές του Λουξεμβούργου πάντα ξεκάθαροι ήταν ως προς αυτό το θέμα. Δεύτερον, έχει τονιστεί ο χαρακτήρας, ο αγοραίος αν θέλετε, γιατί μιλάμε για αγορά δικαιωματών εκπομπών. Αυτή ήταν η εναλλακτική που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ρύθμιση του ζητήματος αυτού. Αυτή την έννοια λοιπόν, σημειώνεται πως μια αγορά δεν μπορεί να αλλοιώνεται, δεν μπορεί να ε, τροποποιείται με κανόνες που έρχονται από τις ε, δημόσιες αρχές. Αυτή λοιπόν η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος θα ήταν ένα παράδειγμα της τροποποίησης της αλλαγής των κανόνων ανταγωνισμού από τον κανόνα του παιχνιδιού από τις δημόσιες αρχές. Εγώ θέλω να πω ότι πρόκειται για μια περίεργη αγορά, αν θέλετε. Είναι λίγο τεχνητή δηλαδή αυτή η αγορά. Και τώρα υπάρχει κάτι ακόμη. Είναι μια περίεργη, γιατί λέω, μια περίεργη αγορά, διότι ουσιαστικά δορίζονται τα προϊόντα. Εγώ δεν γνωρίζω να δορίζονται προϊόντα σε καμιά άλλη αγορά. Επομένω, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το ιδιόμορφο, το ιδιαίτερο και δεν ε, μας παραξενεύει βέβαια ταυτόχρονα ότι ναι με λειτουργεί ω αγορά, αλλά όχι ω μια παραδοσιακή αγορά. Και επειδή πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, βλέπουμε τον Άγιο Βασίλη που έρχεται με τα δώρα. Μάλλον με αυτό μοιάζει πιο πολύ παρά με μια αγορά. Τρίτον, πολύ σωστά πιστεύω και με ε, λογική έχει τονιστεί το θέμα των ε, κρατικών ενισχύσεων λόγω της άξονα των τιμών. Κράτη που έχουν βέβαια χρήματα γιατί κάποια άλλα δεν έχουν θα μπορούσαν να στηρίξουν κάποιες επιχειρήσεις, κάποιους τομείς για να ανεβούν οι τιμές παραλαμβάνω. Αυτό είναι πιθανό και εφικτό. Αυτές οι ενισχύσεις όμως από τα κράτη θα πρέπει να εγγράφονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων που ρυθμίζονται πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και δεν μπορεί ελαφρά τη καρδιά να γίνεται αυτό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως γνωρίζουμε, δηλαδή να δίνει ένα κράτος ενισχύσει έτσι. Επομένω είμαστε υπέρ της πρότασης της Κομισιόν και είχα πει στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων ότι η πρόταση της Κομισιόν πρέπει να θεωρείται ως κάτι έκτακτο. Δηλαδή, έχουμε να δράσουμε απέναντι σε μια οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση πολύ μεγάλης ε, σπουδαιότητας. Επομένως, η Κομισιόν ενεργεί ε, με αυτό το γνώμονα, έχοντας ε, υπόψη στην κρίση και υιοθετώντα έκτακτα μέτρα. Ένα άλλο θέμα θα μπορούσε να είναι η ανάλυση όλων των ζητημάτων τη αγορά, των δικαιωμάτων εκπομπών για το μέλλον. Να δούμε δηλαδή τι μπορεί να γίνει, τι έχει λειτουργήσει σωστά, τι δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Εγώ νομίζω ότι και αυτή είναι μια δική μα αποστολή, μια αποστολή για το Κοινοβούλιο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Η Κομισιόν πρέπει να πω ότι ήδη έχει κάνει μια σημαντική προσπάθεια για να διευκρινίσει, να διαφωτίσει την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών όπως την εννοεί έχει δημοσιεύσει μια πληρέστατη έκθεση για την κατάσταση αγοράς άνθρακα με έξι διαφορετικές εναλλακτικέ για την οργάνωση όλων αυτών. Άρα είναι ένα ζήτημα για το μέλλον, πράγματι, που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε. Και επαναλαμβάνω, όπω είπα και πριν, να δούμε τι λειτουργήσε σωστά, τι λειτουργήσε άσχημα και να επιφέρουμε αλλαγέ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαφορετική συγκυρία που την χαρακτήρισα έκτακτη. Και θέλω να επισημάνω ένα συγκεκριμένο στοιχείο ε, της νομοθεσίας για, ε, για τον πληστηριασμό των ε, δικαιωμάτων εκπομπών. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να το συζητούμε, γιατί δεν εξαντλείται το αντίθετο, το ζήτημα αυτό, το ΣΕΦ και σίγουρα πρέπει πρέπει να έχουμε υπόθεση και τα νομικά μέσα που έχουμε εκπονήσει μέχρι τώρα, τα νομικά μέσα που έχουμε εκπονήσει, παραλαμβάνω, μέχρι στιγμής και κυρίως την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση που θα πρέπει και αυτή να εμπνεύσει και άλλε μεταγενέστερες δράσεις. Δηλαδή να ξέρουμε ότι εμείς δρούμε ω νομοθέτε σε, σε μια συνέχεια. <clears throat> δεν πρέπει να υπάρχουν ρογμές, δεν μπορεί να υπάρχουν αντιφάσεις, ιδίως αυτές τις πάρα πολύ ε, ορατές που βλέπουμε και φανταχτέρες αν θέλετε. Δεν πρέπει να τις βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παραπονεθώ για την μετάφραση. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ε, να υπάρχουν, ε, να βρεθούν διερμηνείς, αλλά μια και έχω συγκεκριμένα αρμοδιότητες, συγκεκριμένα καθήκοντα, ε, για μια και είμαι σκιώδης εισηγήτρια, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχω, να έχω να μπορώ να μιλάω στη γλώσσα μου. Λοιπόν, οι πληστηριασμοί δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίων είναι σημαντικοί. Το πρόβλημα είναι ο μηχανισμός αυτός σε τι αποσκοπεί. Άλλοι λένε να μαζέψουν χρήματα, άλλοι λένε να μειωθούν οι εκπομπές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ισχύει το δεύτερο. Ο, ο, οι πληστηριασμοί αυτοί έχουν σαν βασικό στόχο να μειώσουν τις εκπομπές. Όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και την οξυσία να κάνει κάποιες αλλαγές. Αλλά θα πρέπει να τεθούν ε, σε, ενέργεια μόνο εάν δούμε ότι δεν σεβόμαστε τους στόχους του 2020 αυτό και όχι οι τιμές. Οι τιμές είναι ένα θέμα αγοράς. Λοιπόν, εάν η Κομισιόν μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες ότι δεν θα σεβαστούμε τους στόχους του 2020 για τις εκπομπές διοξυδίου του άνθρακα, τότε, τότε θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις σχετικά με τους πλησιρισμούς, εκτός βέβαια αν υπάρχουν διαρροές διοξιδίου του άνθρακα, που εκεί υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είπε και ο εισηγητής. Μπορούμε να δεχτούμε κάποια ad hoc απόφαση, μόνο όμως για βραχυπρόθεσμα μέτρα και με ιδιαίτερους περιορισμούς, διότι εμείς λαμβάνουμε αποφάσεις, όπως είπε και ο εισηγητής. Μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε για την ευελιξία του μηχανισμού αυτού, διότι το μηχανισμός δεν είναι ευέλικτος και εδώ υποστηρίζω απόλυτα την συζήτηση που γίνεται για διαδροτικές αλλαγές του μηχανισμού αυτού που θα μας δώσουν περισσότερο, να εξασφαλίσουν περισσότερη ευελιξία ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν και σταθερότητα στους επενδυτές. Χτες ε, έγινε μια συζήτηση και για τον, το σύστημα αυτό των πληστηριασμών, ακόμα και στην Επιτροπή ΕΜΒΗ δεν εξασφαλίζουν υποστήριξη, αμέριστη υποξήση στην Κομισιόν. Και εκεί ο εισηγητή ε, έθεσε κάποιους περιορισμούς για το πόσε φορέ ε, μπορεί να αλλάξει το σύστημα. Τέλο πάντων, συζητιώνται οι προποθέσει. Τέλο πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το επανεξετάσουμε πιο σοβαρά το θέμα των ε, πληστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Μέρκης. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, κύριο Σώσα για την πάρα πολύ καλή επισκόπηση αυτού του, ε, αυτής της πολύ σημαντική πρόταση για την δρομολόγηση αυτής της αγοράς. Σύμφωνο και με σας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί αυτή η αγορά. Και αυτό είναι σαφές ε, και ακόμη περισσότερο λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρέπει λοιπόν να παρέμβουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν δουλεύει. Είναι μια ιδιαίτερη αγορά, δεν είναι μια συνήθις αγορά. Είναι μια ιδιαίτερη αγορά στην οποία, όπως ε, είπατε κι εσείς, ε, έχουμε δώσει πολλά δωράκια. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συνήθως σε μια λειτουργούσα αγορά. Υποστηρίζω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι πρέπει να παρέμβουμε και πιστεύω ότι το backloading είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να παρέμβουμε αμέσως. Συμφωνώ όμως και το, με τον συνάδελφο Κρότε στην ε, ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι το δικαίωμα της ε, παρέμβασης δεν πρέπει να μας κάνει τόσο χαρούμενους ώστε να παρεμβαίνουμε συνεχώς πρέπει με πολύ διαρθρωμένο τρόπο να παρέμβουμε για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε το σύστημα αν χρειαστεί, αλλά όχι πέρα από αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ασφάλεια, γιατί κάθε αγορά χρειάζεται σταθερότητα και κάποιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πρέπει όμως να δράσουμε αμέσως Αναμένω εναγωνίως συζήτηση για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Έχουμε κάποια επιχειρήματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσω, γιατί ακούγονται πολλά όσον αφορά τις ε, απαιτητικές ενέργεια ε, βιομηχανίες που μπορεί να πληγούν ε, λόγω του ε, συστήματος εμπορίας αερίων. Υποφέρουν και θα εξακολουθήσουν να υποφέρουν μετά το 2013 δεν θα υπάρξει ιδιαίτερος αντίκτυπος για αυτές λόγω του μέτρου backloading. Για παράδειγμα, η χαλιβουργία, και μάλιστα μόλις ε, εγκρίναμε ψήφισμα γι' αυτό, δεν μπορούν να μειώσουν κι άλλο τις εκπομπές τους. Ε, έδειξε μία μελέτη ότι πέρα από τη χαλιβουργία, ότι μπορούμε ακόμα 16 ε, έως 32% να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ποιο ακριβώς τομέα θα στοχεύσουμε. Κατά πόσο πρέπει να παρέμβουμε σε μία αγορά και αν είναι φυσιολογικό αυτό, ναι είναι και το έχουμε δει και σε άλλες αγορές. Νομίζω ότι η παρέμβαση υπέρ της ε, ε, ζήτησης ε, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Για να είμαι λοιπόν πολύ σύντομη, αναφέρθηκατε στα βασικά στοιχεία της Άποψη του κυρίου Γκρότε. Συμφωνώ με τα βασικά στοιχεία της άποψής του και κυρίως με το ότι πρέπει να επιτρέψουμε ένα μόνο backloading. Η κυρία Χάλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόσα Βάγνερ, ε, πάρα πολύ μάλιστα, για την έκθεσή του. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό πρέπει να επιβεβαιώσουμε μία νομική βάση, να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Ούτως ή άλλως όμως η αλλω ομως Επιτροπή έχει κάνει ήδη τις προσαρμογές ε, στο ε, πρόγραμμα εμπορίας, στο σύστημα εμπορία αερίων και κανένας ε, δεν ασχολήθηκε με αυτό. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία αμφισβήτηση αυτού που θέλουμε να επιτύχουμε Είπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει ασφάλεια δικαίου και αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε κι εμείς είναι ένας μηχανισμός αγοράς. Όντως είναι ένας μηχανισμός αγοράς, αλλά όπως είδαμε και με τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές, μερικές φορές οι, αγορές χρειάζονται ρυθμίσει, σε μερικές ε, περιπτώσεις ε, δεν λειτουργούν όπως πρέπει και γι' αυτό πρέπει να παρέμβουμε για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία τους. Αυτό έγινε και στην προκείμενη περίπτωση με το σύστημα εμπορίας αερίων. Διάφοροι παράγοντες συνετέλεσαν, ιδιαίτερα η οικονομική κρίση αλλά και άλλα πράγματα. Ε, που έχουν μειώσει την τιμή του άνθρακα σε πολύ πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που αναμενόταν. Ε, είναι μια πολύ μετριοπαθής αυτή η ε, δυνατότητα του backloading για το ποσό που προτείνεται. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επανέλθει με πιο μακροπρόθεσμες και στρατηγικές λύσεις, γιατί συμφωνώ και με τη συνάδελφο που είπε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την επίτευξη των στόχων για το 2020, αλλά και για το 2050. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους δεύτερους στόχους ε, αν δεν επιδοτήσουμε άμεσα πολύ τον κλάδο. Αλλιώς, αλλιώς πρέπει να δώσουμε κίνητρα για τη μείωση του άνθρακα και με, την, με, τις, με το επίπεδο των τιμών του άνθρακα αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει το κίνητρο να επενδύσει σε ε, χαμηλό ε, ε, άνθρακα. Αντιθέτως, ε, ε, σκέφτονται μήπως θα έπρεπε να επιστρέψουν στο χάλιβα Έχουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους για τον άνθρακα μέχρι το 2050. Δεν θα μπορέσουμε όμως να τους επιτύχουμε αν δεν αλλάξουμε το σύστημα εμπορίας αερίων και ε, αν δεν επιτρέψουμε στην αγορά να λειτουργήσει σωστά. Θα ήθελα να ζητήσω Ας μην το κάνουμε ευχολόγιο αυτό το πράγμα που έχουμε μπροστά μα. καλύτερα να το ε, διατηρήσουμε απλό. Θέλουμε να επιτύχουμε την ασφάλεια δικαίου, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει αυτό το backloading που θέλει. Ευχαριστώ. Η Πιλάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχά να σε να ευχαριστήσω τον Σάλφο Σαβάγκνερ για την παρουσίαση και τις προτάσεις του. Λοιπόν, ξεκινάμε ότι έχει πολλές και καλές προθέσεις κομισιών. Και η Επίτροπος που είναι πολύ θαραλέα. Γιατί πραγματικά τέτοια αντιμέτωπη με σθένος σε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την του κλίματος. Όλα αυτά τα αναγνωρίζουμε. Όμως εδώ, πολύ απλά, μας επηρεάζει νομίζω αυτό το πολύπλοκο πράγμα που έχει ε, ως χαρακτηριστικό η, δημιουργία, η τεχνητή δημιουργία μιας αγοράς. Όταν δημιουργούμε μια τεχνητή αγορά υπάρχουν, προκύπτουν καταστάσεις όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν τα προβλήματα. Όταν είχαμε οικονομική ανάπτυξη, αυτό συγκάλυψε πολλά πράγματα όχι μόνο σε σχέση με την τεχνητή αγορά, αλλά και πάρα πολλές άλλες πτυχές πραγματικότητας ε, των οικονομιών των πολλών, των περισσότερων χωρών της ε, Ένωσης. Ενώ βλέπαμε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση Όταν όμως έχουμε την πλημμυρίδα, όταν έχουμε την άποτη, βλέπουμε ποιος είναι γυμνός όταν κατεβαίνουν τα νερά. Και σε φόρα το είτε. Στον έπεσε λοιπόν, όταν η συγκύρια πια δεν ήταν καλή, είδαμε τα προβλήματα αυτής της αγοράς, που δεν με μια τεχνητή αγορά. Πώς αντιμετωπίζει λοιπόν μια αγορά, μια κατάσταση κρίσης. Είναι διαφορετικές απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς. Μπορεί να δώσει κίνητρα, φορολογικά για παράδειγμα αλλά όχι να παρέμβει άμεσα στη διαμόρφωση των τιμών. Θα μπορούσε να προτείνει νομοθεσία για να προωθήσει περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και ούτω καθεξής. Εδώ όμως δεν γίνεται αυτό και ρυθμίζουμε απευθεία τις τιμές. Αυτό σχετίζεται με τον, τεχνικό, με τον τεχνητό συγγνώμη, αυτό χαρακτήρα της αγοράς αυτής. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται αυτό γιατί δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι για τη μείωση εκπομπών το 2020. Η ίδια Κομισιόν αναγνωρίζει ότι πράγματι είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε τους στόχους. Γιατί γίνεται. Γίνεται για να υπάρξει ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου. Το είπε και η Φιώνα Χόλ. Ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές και πέραν του 2020. Για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια δικαίου όμως, οι τιμές αποσυνδέονται από το προϊόν που είναι τα δικαιώματα εκπομπών. Δεν νομίζω προσωπικά ότι αυτό θα λειτουργήσει τελικά. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια βιομηχανία που θα παράγει. Όχι μόνο σε κάποιες χώρες της Ένωσης. Αν θέλουμε να έχει νόημα και αν θέλουμε αυτά τα δικαιώματα εκπομπών και οι τιμές τους και να μπορεί να γίνει η αγορά τους είπε πως Μέρκης για τις βιομηχανίες τις ενεργοβόρες. Ότι πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικές και μπορούν, γιατί μπορούν να πάρουν κάποιες ενισχύσεις. Πράγματι, είναι αναγνωρισμένες από το 2013 και μετά αυτές οι άμεσες ενισχύσεις. Εντάξει, πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να καταβληθούν ενισχύσεις αυτές και υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορούν να δώσουν τις ενισχύσεις αυτές, τις άμεσες αυτές ενισχύσεις στις ε, ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και αυτό αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις εν λόγω επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και να έχει, εγώ νομίζω ότι αν τελικά προχωρήσει αυτό, ξεκολουθούν να υπάρχουν ζητήματα και κάποια όρια, και, ε, ε, που θα πρέπει να μπουν. Δηλαδή, πώς η Κομισιόν, αφού του τεθεί σε αυτό το μέτρο, πώς η Κομισιόν λοιπόν θα πανησαγάγει και θα επαναθεσπίσει τα δικαιώματα εκπομπών που είχαν αποσυρθεί. Πώς θα γίνει αυτό γραμμικά και προοδευτικά, βαθμιαία και κάποια άλλα θέματα. Όλα αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκύπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάποια κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ε, προστασίας του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν αυτό τον μηχανισμό. Αλλά αυτό όμως δεν ξέρω αν είναι σωστό να το ενθαρρύνουμε. Ε, σαν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε υιοθετήσει πολλούς κανόνες για τον περιορισμό των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου και πιο συγκεκριμένα διοξιδίου του άνθρακα και πολλές χώρες στη Γερμανία, η Ισπανία έχουν χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλουμε να τιμωρήσουμε την βιομηχανία. Πρώτα τους αναγκαιάζουμε να, υιοθε... να επενδύσουν σε τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος. Καλό είναι αυτό είναι. Ε, θέτουμε στόχους για περιορισμούς των εκπομπών, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ε, τώρα ε, τιμωρούμε την βιομηχανία για μια καινούργια φορά μέσω αυτών των οπλιστηριασμών. Είναι μια πολιτική την οποία να προτείνει η Κομισιό, την οποία δεν καταλαβαίνω, φίλο να ομολογήσω. Και εάν, όπως είπε ο συνάδελφος, επιτρέψουμε να συνεχίσει αυτό και να γίνει μία φορά, τότε δεν πειράζει. Αλλά αυτό δεν ισχύει, διότι και μία φορά να εφαρμοστεί, θα, η Κομισιόν θα το συνεχίσει και θα επιτρέψει να γίνεται ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δάλκουρα Σε Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για να πω κάτι στον καθηγητή Σώσα. Μια νομοθετική πρόταση με ένα μόνο άρθρο. Δεν νομίζω ότι σας κόστησε και πολλή δουλειά. Ε, και δεν είναι και... Δεν, δεν τη χάνει και ομοφωνίας. Λοιπόν, έχετε πει σημαντικά πράγματα και θέλω και εγώ να πω ότι ναι, μεν συμφωνώ με τα περισσότερα, αλλά ε, με ένα από αυτά διαφωνώ και χαίρομαι, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ βαρετή και μονότονη η σχέση μας. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι εστιάζεται σε μια πτυχή που νομίζω πρέπει να την αναθεωρήσουμε, δηλαδή η αγορά δικαιώματα μπορεί να δεν είναι αγορά. Η κυρία Μέρκης είπε είναι μια ιδιαίτερη αγορά, μια ειδική αγορά. Αυτό είναι ένας ωραίος εφημισμός για να πούμε ότι δεν είναι αγορά. Πολύ απλά. Δεν είναι αγορά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μία εφεύρεση. Είναι ένα τεχνητό ε, δημιούργημα ώστε τελικά να δημιουργήσει δημόσια εξουσία μία αγορά που δεν υπάρχει. Γιατί φυσικά και αυθόρμητα δεν ε, απαντά στον κόσμο κάτι τέτοιο για να μπορεί να, πληστη... να βγαίνουν στο πληστηριασμό αυτά τα δικαιώματα και αυτή η αγορά η τεχνητή τελικά λέμε ότι θα εξελιχθεί κατά τρόπο που θα μας στάσει σε μια ευτυχή ε, κατάσταση που θα μειωθούν οι κόμπες. Μα δεν γίνεται έτσι. Μια αγορά αφού δεν είναι αγορά πώς θα λειτουργεί σαν αγορά. Και πράγματι είδαμε ότι λόγω της κρίσης ε, και άλλων πολλών θεμάτων μειώθηκαν οι τιμές, πέσαν οι τιμές. Και το μόνο που μας προτείνει τώρα η Κομισιόν είναι να παρέμβει σε αυτή την υποτιθέμενη αγορά, επαναλαμβάνω, να μας αποδείξει ότι είναι ενώ δεν είναι και να δημιουργήσει τελικά και νέα προβλήματα. Για παράδειγμα, επειδή μνώνεται σημαντικά η ανταγωνιστικότητα βιομηχανικών κλάδων, πάρα πολύ σημαντικών, στρατηγικών κλάδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, για να δούμε και το γενικότερο πλαίσιο. Υπάρχουν χώρες που εκπέμπουν πολλές εκπομπές, ε, όπως είναι ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ρωσία. Και κάνουν πίσω. Υπαναχωρούν και δεν δέχονται την παράταση του Κιώτο. Το είδαμε και στην Τόχα. Επιμένουμε εμείς όμως να, μας, αυτό Το πόδι μας πάνε όλοι από την άλλη κατεύθυνση και εμείς θα μπορούσαμε ε, τελικά να καταστραφούμε ενδόξως. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό. Μπορεί να έχει και μία αξία αυτό, αλλά δεν ξέρω τι ικανοποίηση προσφέρει. Τέλος πάντων. Επομένως, λέω, δεν είναι αγορά. Πώς θα παρέμβει κάποιος σε μια αγορά που δεν είναι αγορά, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζουμε τα λάθη. Και εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Πίπερ σωστά είπε ότι καλό θα ήταν να το ξεχάσουμε αυτό το θέμα. Βέβαια, για να αφήσω και έτσι μια πόρτα ανοιχτή, θα μπορούσε, θα μπορούσε να εξεταστεί ένα τέτοιο μέτρο με δύο όμως προϋποθέσεις, με δύο όρους. Πρώτον, εάν δεν εκπληρώνονται οι στόχοι, που δεν συμβαίνει γιατί τους εκπληρώνουμε τους στόχους και δεύτερον, να μην πληγεί σημαντικά η ανταγωνιστικότητα των ε, κλάδων αυτών και των ιστών. Με αυτές τις προφυλάξεις τις δύο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να παρέμβει η Κομισιόν σε αυτή τη μία αγορά. Αλλά όπως είναι τα πράγματα και όπως είναι έτσι η έκθεση, νομίζω το μόνο στο οποίο θα οδηγήσει θα είναι νέες καταστροφές. Καθηγητά Σώσα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό σας θαυμάζουμε Τα διανοητικά λάθη οδηγούν σε σοβαρά λάθη άλλου τύπου. Και στην προκειμένη περίπτωση η Κομισιόν ξεκινά από ένα σοβαρό διανοητικό λάθος και μας βάζει σε αυτό το χάος που πρέπει τώρα εμείς να το ξεμπερδέψουμε. Ευχαριστώ, η συνάδελφος κυρία Κόρολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπεύθυνη για τη θέση της, ε, του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα ήθελα συνεπώς να κάνω κάποια σχόλια για το θέμα αυτό. Άκουσα πολλούς συναδέλφους να λένε ότι πρόκειται για τη μείωση των εκπομπών αερίων και για την εξασφάλιση ότι θα, παραμένουμε, θα παραμείνουμε στο σωστό δρόμο. Να σας πω κάτι όμως. Το σύστημα εμπορίας αερίων ούτως ή άλλως από μόνο του μειώνει ε, τους, ε, τις εκπομπές αερίων αυτομάτως. Δεν χρειάζεται να αυξήσουμε λοιπόν ε, ε τις, ε, τιμές, τις τιμές του ηλεκτρισμού για να το κάνουμε, για να το πετύχουμε αυτό. Δεύτερον, μείωση των εκπομπών της παραγωγής. Περί αυτού πρόκειται. Όμως, βάσει του Κιώτο, αυξήσαμε εμείς τις εκπομπές αερίων μας. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατανάλωση στην Ευρώπη. Αν δούμε λοιπόν τις συνολικές μας εκπομπές αερίων και τις κατανάλωσης, οι στατιστικές ε, του Διεθνούς Εμπορίου δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει τις εκπομπές αερίων κατά τη διάρκεια των μέτρων για το κλίμα. Και το κάνουμε μάλιστα μέσω του ETS. Ε, ε, Κάνω εξωτερική ανάθεση του κλάδου και των εκπομπών μας εκτός Ευρωπα... Ευρώπης και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο πρέπει να διασφαλίσουμε αυτό το ETS σε τέτοιο βαθμό για λόγους ε, πολιτικής υπερηφάνειας, ας πούμε. Θέλουμε να το σώσουμε γιατί εμείς το δημιουργήσαμε και θέλουμε να προστατεύσουμε τη φήμη του. Θα ήθελα να μου πείτε πραγματικά, εμένα με ενδιαφέρει το να μειώσουμε τις εκπομπές μας, αλλά γιατί θέλουμε τόσο πολύ να σώσουμε το ETS. Ε Όσον αφορά λοιπόν τώρα ειδικά τους πληστηριασμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει στους κανόνες του ETS, ε ακόμη και αν είναι κάποιο είδους ελιγμός, ε, το κόστος ενέργειας θα εξακολουθήσει να αυξάνεται και συγκεκριμένα ο άνθρακας και σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στη μείωση των εκπομπών αερίων ε, ε, εις βάρος όλων όσων ήθελε να εξυπηρετήσει αυτό το σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζουμε ως αντάλλαγμα την ανταγωνιστικότητα της θέσης απασχόλησης. Ε, επίσης, ε, ε, πλήττεται και η αξιοπιστία του ETS ως, ως μηχανισμού της αγοράς. Κάτι το οποίο έχει συμβεί ήδη πιστεύω σε μεγάλο βαθμό έχει προβλεφθεί ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρισμού θα αυξηθούν ε, πάνω από 3%, δηλαδή 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω αυτών των ε, προγραμμάτων και πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτή η αλλαγή των κανόνων των πληστηριασμών συνάδει με την ε, τρέχουσα νομοθεσία του ETS. Το άρθρο 9 λέει κανένα backloading των ε, μεταφορών από τη μία χρονιά στην άλλη, θέτει πολύ συγκεκριμένους όρους ε, ε, για τα δικαιώματα των, των εκπομπών αερίων, ούτως ή άλλως, οπότε... Δεν καταλαβαίνω γιατί παρεμβαίνουμε σε τέτοιο βαθμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στούρμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί κάποιοι λένε ότι έχουμε διανοητικά χρεοκοπήσει και ίσως θα έπρεπε να μετράμε τις επιδόσεις ο ένας του άλλου, ίσως. Όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, Υπάρχει ένα, ε, τα στοιχεία αυτά ε, μας τα δίνει ένα λόμπι γερμανικό που, αφορού, που αφορά τις σχέσεις και αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στις εκπομπές, ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι οι μελέτες που έχουν γίνει και οι στόχοι της Ευρώπης του 2020 παρουσιάστηκαν το 2007. Και όταν έχουμε 20% ανανεώσιμες και 20% μείωση ε, εκπομπών του αερίου, τότε πασπερισσεύει, αν θέλετε, ε, κάποιες μας περισσεύουν κάποιες ε, εκπομπές και ε, ούτως ή άλλως το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι τιμές και θα παραμείνουν μειωμένες οι τιμές οφείλεται στο γεγονός ότι η Κομισιό με βάση τις γνώσεις που είχε το 2007 για λόγους που ποτέ δεν κατανόησε παρουσίαση ένα πακέτο 20-20-20%. Ενώ για να υπάρχει ένα κάποιο ενδιαφέρον στην αγορά ε, πληστηριασμών θα έπρεπε να είχαμε 20-20-40 ή 35 ε, με 40% μείωση μέχρι το 2020. Ε, θέλουμε επομένω ε, να είμαστε ιστορικά και διανοητικά σωστοί αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ιστορία και αυτό το βασικό πρόβλημα. Επομένως, ένας τρόπος για να διορθώσουμε το λάθος είναι να έχουμε 20%, 20 ε, το 2020. Το άλλο επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του καθεστώτος και του backloading θα προωθήσει την βιομηχανία. Μήπως να διαβάσετε, να διαβάσετε τις ε, ομιλίες σας το 2007. Ήμουν εκεί παρούσα και τότε ήσασταν παρόν συγγνώμη, και ήσασταν ε, πολύ πιο ε, αισιόδοξοι για το σύστημα αυτό των πληστηριασμών. Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω πώς βλέπετε με τέτοιο διαφορετικό τα πράγματα, με τόσο διαφορετικό τρόπο τα πράγματα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Για 10 δευτερόλεπτα εστιάστε την προσοχή σας. Όταν έχουμε 4 με 5 ευρώ τον τόνο το, το σύστημα πληροφοριασμών, πώς μπορεί κάποιος κάτι που έχει τόσο χαμηλή τιμή να αποτελέσει ένα κίνητρο για την ε, ε, ε, αλλαγή της βιομηχανικής θάλασσας της Ευρώπης. Και ήδη με την ανακοίνωση της Κομισιόν το 2007-2008, όταν μιλούσαμε για τη μεσα τονο ανατόνο 15-20, υπήρχαν πολλά οικονομετρικά μοντέλα που έλεγαν ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε τιμή στη μέσα 15-30 αρκεί να υπάρχει αντιστάθμιση. Και ας ολοκληρώσω ε, το επιχείρημά μου, πως σας παρακαλώ. Αυτό κανείς, κανείς δεν, δεν, από εσά δεν ανέφερε ότι υπάρχει αντιστάθμιση, ε, ότι υπάρχουν μάλλον αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται, διότι οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις οι ε, εντατικής ενέργειας εφαρμόζουν την καλύτερη δυνατή τεχνολογία και μετά η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού δέχτηκε μια παγωμένες ε, τιμές μέσω αυτού του συστήματος, του μηχανισμού. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μία τιμή φθορίου ε, διοξείδου του άνθρακα και το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανά να τελειώσω την ε, πρότασή μου. Το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανά το 10% ε, των εσόδων από το μηχανισμό πληστηριορισμού και αντισταθμίζει τις, ε, και μάλλον αποζημιώνει τις επιχειρήσεις αυτές. Επομένως, τα επιχειρήματά σας δεν είναι σωστά και απλώς ε, ακούτε τα επιχειρήματα ενός λόμπι εταιριών και επιχειρήσεων εντατικής ενέργειας, αν θέλετε, που θέλουν να καταστρέψουν το σύστημα. Ο κύριος Γκέμπελς έχει τον λόγο. Παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που δεν τους άκουσα, αλλά θα ήθελα να απαντήσω στα επιχειρήματα του εξαιρετικού συναδέλφου κύριου Τόμας που λέει ότι επειδή η τιμή των πιστοποιητικών είναι τόσο χαμηλή δεν μπορεί να κάνει κακό, δεν μπορεί να κάνουν κακό. Ο στόχος όμως της Κομισιόν είναι να αυξηθούν τεχνητά οι τιμές και αυτό θα προκαλέσει κακό διότι όπως είπε και ο συνάδελφος Βιντάλ Κουάντρας Είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που πιστεύουν για ένα μέτρο το οποίο δημιούργησαν τα παιδιά, τα αγόρια από το Σικάγο. Αυτό το σύστημα των εκπομπών διαδόθηκε όταν αντιπρόεδρος ήταν ο Αλ Γκόρ, όταν υιοθετήθηκε το πρωτόκολλο του Κιώτο. Όμως όταν ξαναγύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γερουσία ε, στράφει εναντίον του Κιώτο, ομόφωνα. Τώρα η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση λέει ότι καταφέραμε να σώσουμε το Κιώτο. Εμείς όμως μόνοι μας, μόνοι εμείς, το, το Λίχτενστάιν, η Ελβετία, η Κροατία, ε, πιστεύει και η Νορβηγία πιστεύουν σε αυτό το πρωτόκολλο του Κιώτο και σε αυτό το μηχανισμό που ε, ε, αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπικών κινήσεων. Είδατε τι έγινε στην προηγούμενη εβδομάδα στην Γερμανία, στην Deutsche Bank, με την Deutsche Bank. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται κερδοσκοπικές κινήσεις πάνω σε αυτά τα δικαιώματα μόλυνσης. Αγαπητέ Κλοντ, Μπορώ να σου δώσω χιλιάδες παραδείγματα όπου έχουν γίνει κερδοσκοπικές κινήσεις. Εδώ όμως κάνουμε το... Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Ε, γιατί πολλές φορές αυτά τα οποία αποφασίζουμε ε, μας οδηγούν σε ε, καταστάσεις ε, που δεν θέλουμε. Λοιπόν, είμαστε οι μόνοι οι οποίοι εξακολουθούμε να πιστεύουμε αυτό το σύστημα το οποίο εφήβρανε τα αγόρια από το Σικάγο. Και εγώ θα το καταψηφίσω τους ή άλλους. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Σαρτόρη, η τελευταία παρέμβαση από τον κύριο Βιντάλ Κουάντρας. έκανε κάποιες παρατηρήσεις ο πολύ καλός φίλος Κλωτούρνας και θέλω να απαντήσω για σε μερικές από αυτές. Μία μελέτη δεν μπορεί ε, να την ε, απορρίπτουμε. Μπορεί να είναι αυστηρή, να είναι ακριβής, ε, να είναι σωστή, να μην είναι, αλλά όχι να την απορρίπτουμε μία θέση, μία μελέτη αυτής εξ αρχής. Επειδή κάποιος συγκεκριμένο την έχει καταρτήσει. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Εμεί πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεύτερον, λέγεται ότι αυτό είναι ένας ελιγμός από τα λόμπι της βιομηχανία, της ενεργοβόρη βιομηχανία. Με εδώ δεν υπάρχει διαλεκτική αλληλεπίδραση διαφανής μεταξύ νομικών συμφερόντων. Φυσικά και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες επαγρυπνούν για τις θέσεις εργασίας τους, για τα κέρδη τους. Και αυτό έλειπε να μην το έκαναν κιόλα. Αλλά από το να φτάσουμε να λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα είδος ε, συνωμοσία των βιομηχανικών λόμπι, μα εδώ τι προσπίζει ο καθένας από εμάς. Είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε με τιμή και με τη λογική μας, που μας πρέπει να καταλαβαίνουμε κάπως τα πράγματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα αλληλοσεβασμού κινούμαστε και συζητούμε. Και άλλωστε όλοι συνάδελφοι είμαστε. Ένα λεπτό γιατί δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση ίδρο. Λοιπόν, το μόνο πράγμα το οποίο είπα είναι ότι το ότι τότε το, όταν, όταν δημιούργησαν το σύστημα αυτό ήταν το 2007 τον Γενάρη του 2007 η Κομισιό είχε θέσει κάποιους στόχους. Τώρα, κύριε Γκέμπελος, γιατί η Κομισιό ε, δέχτηκε και προτείνει αυτό το backloading και ποια είναι ο αντίκτυπος της τιμής. Από τον ε, Γενάρη θα έχουμε ευρωπαϊκό σύστημα και όχι εθνικά συστήματα. Χωρίς το backloading οι εμπειρογνώμονες μας λένε ότι η τιμή θα πάει στο μηδέν. Ναι, αλλά εσύ θα χαρείς γι' αυτό. Θέλει να καταστρέψεις το σύστημα. Βέβαια, είσαι ο μόνος, ένα από τους λίγους που το λένε ειλικρινά. Και αυτοί που είναι κατά του backloading ή θέλουν να καταστρέψουν το σύστημα. Κάποιες βιομηχανίες στην Ευρώπη θέλουν να καταστρέψουν το σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα, αλλά στις 6 έχουμε τους ε, συντονιστές. Κύριε Γκέμπελς, ε, τι να σας πω... Μετά θα είναι η συζήτηση ανεξέλεγκτη. Υπάρχει η Κομισιόν Σούζα Βάγνερ, και μετά είναι οι συντονιστέ. Τώρα, αν θεωρείτε ότι θέλετε οπωσδήποτε να παρέμβετε για 30 δευτερόλεπτα, έχετε το λόγο. Απλώ και μόνο να υπενθυμίσω ότι οι συνολικές εκπομπές Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 10% των σφαιρικών εκπομπών. Κάτω από το 11%. Και όλοι που όσες χώρες εφαρμόζουν το σύστημα Κιώτο, στο σύνολο μαζί έχουν 15%. Εάν καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε 15 των εκπομπών, τι θα γίνει? Θα μειωθεί η συνεισφορά μας, αλλά όχι όμως η συνολική, το συνολικό ποσό, η ποσότητα των εκπομπών, διότι οι, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να μολύνουν. Καλώς, ε, η Κομισιόν έχει το λόγο. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Κομισιόν, Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι όντως για την πρόταση αυτή ανταποκρίνεται σε μία έκκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την οδηγία ενεργικής αποδοτικότητας που ολοκληρώθηκε ε, το καλοκαίρι. Ε, γι' αυτό ζητήθηκε η αναθεώρηση και γι' αυτό ακριβώς υποβάλαμε την ε, σχετική πρόταση. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε μία έκκληση προς την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για πιο διαρθρωμένα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση του ETS και γι' αυτό λοιπόν ανταποκρίθηκε ε, μέσω της έκθεσης ε, της αγοράς του άνθρακα και ε, υπέβαλε και κάποια στοιχεία σε σχέση με κάποια μέτρα που μπορούμε να ακολουθήσουμε μακροπρόθεσμα. Να υπενθυμίσω τη λογική πίσω από αυτήν την πρόταση για να υπάρξει επιπλέον ασφάλεια δικαίου για την αλλαγή των δικαιωμάτων είναι η οικονομική κρίση, κάτι το οποίο ήταν απρόβλεπτο ακόμη και όταν αποφασίσαμε το, στο τέλος του 2008 το ε, πακέτο για το κλίμα. Είναι μια εντελώς εξαιρετική κατάσταση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να αρχίσει να παρεμβαίνει με συστηματικό τρόπο στην αγορά. Είπαμε αντιθέτω ότι θα γίνει μόνο σε ε, εξαιρετικές περιπτώσεις όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ισχύει. Θα ήθελα να υπενθυμίσω λοιπόν στα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου ότι υπήρξε ήδη μια αλλαγή μια φορά το 2011 και ότι τότε ε, θεωρήθηκε από τους δύο εμπλεγόμενους φορείς που ζητούσαν αυτήν την αλλαγή ε, να ζητηθεί υπόψη κατ' εξαίρεση κατάσταση που αφορούσε τη μετάβαση από την τρέχουσα φάση 2 στη φάση 3. Όλε, όλα τα δικαιώματα εμπορίας ε, θα τίθενται σε πληστηριασμό και θεώρησαν τότε ότι θα, θα δημιουργούσε τεράστια αύξηση τιμών και γι' αυτό ακριβώς τότε συμφωνήθηκε να αρχίσει το 2012 η φάση 3 των πληστηριασμών και αυτό άρχισε. Το Νοέμβριο λοιπόν του 2012 ήδη ξεκινήσαμε ε, με την πρόταση αυτή. Είναι κάτι το οποίο εξετάστηκε και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και εγκρίθηκε πλήρως. Ε, θέλουμε λοιπόν επιπλέον ασφάλεια δικαίου για την αγορά. Θέλω να, να τονίσω όμως επίσης ε, ότι η επιπλέον... Ε, 900 πλέον 900 εκατομμύρια ε, δικαιωμάτων πάλι θα τεθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή ε, αποφασιστεί ότι υπάρχει δυνατότητα της συναπόφασης για αυτό το τομέα που είναι η αναθεώρηση των του πληστηριασμού των δικαιωμάτων. Και τέλος, θα ήθελα να απαντήσω στα σχόλια που έγιναν όσον αφορά τον αντίκτυπο στον κλάδο και στις τιμές του ηλεκτρισμού. Να τονίσω καταρχάς ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο πώς θα επηρεαστούν οι τιμές. Αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι ένα μέτρο διαχείρισης ε, ε, της ε, προσφοράς. Ε, είναι κάτι το οποίο ήδη αναφέρεται στην επιτρο... στον κανονισμό της Επιτροπής, ότι θα ξανατεθούν στην αγορά αυτά τα δικαιώματα το 2019-2020. Άλλωστε μπορεί να μειωθούν και οι τιμές γιατί υπήρχε ήδη μια τιμολόγηση πριν αρχίσει να ισχύει το backloading. Υπάρχει περίπτωση να είναι μετριασμένη αύξηση των τιμών, τέλος πάντων, ε, σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι θεωρούσαμε όταν εγκρίναμε το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα. Αν χρειάζεται περαιτέρω ε, πληστηριασμό, αν, χρειάζεται, ε, αν, υπάρξει περαιτέρω, αν υπάρξουν περαιτέρω έσοδα, τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν για την ε, αντιστάθμιση ορισμένων ε, προβλημάτων του μηχανισμού για των ενεργειών ε, των κλάβων που είναι πολύ απαιτητικοί σε ενέργεια, για παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. τον λόγο τον έχει ο κύριος Σούζα Βάγνερ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μίλησαν και τους και τους αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους που βοήθησαν να απλουστεύσουμε λίγο, να ξεμπεριλδέψουμε αυτό το πολύπλοκο ζήτημα και ευτυχώς που ξεκινάμε από την ιδέα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια τεχνητή αγορά. Ο φίλος Αλέχο την προηγούμενη φορά που τα συζητήσαμε λίγο ότι είναι αγορά. Τώρα όλοι δεχόμαστε ότι δεν είναι αγορά. Είναι μια τεχνητή αγορά. Είπα, δεν ήσασταν εδώ, αλλά το λέω, ότι είναι περίεργη αγορά γιατί δορίζονται τα προϊόντα. Και δεν νομίζω ότι σε κάποια άλλη αγορά δορίζονται προϊόντα. Είπα όμως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν έχουμε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές που υπάρχουν παρεμβάσεις εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας χρηματοοικονομικών προϊόντων λόγω της μαζικής παρέμβασης από τη δημόσια εξουσία, τη δημόσια χρήμα. Πώς εδώ θα μπορέσουμε αυτό να το αποφύγουμε. Άρα μπορεί να υπάρχει παρέμβαση από την αγορά. Αλλά με βάση αυτό το μέτρο που προτείνει η Κομισιόν τώρα. Και τέλος, να πω ότι σε ό,τι αφορά την επιδείνωση της αγωνιστικότητας, εδώ παρουσιάστηκαν εκθέσει κάποιων επιχειρήσεων. Τώρα είναι λόμπι, δεν είναι. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω για εκθέσεις από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Λόγω των πεπιθήσεων και των πολιτικών αλλά και των σπουδών μου νομίζω ότι οι κυβερνήσεις εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον μέσα στο δημοκρατικό σύστημα. Και αυτό που μα λένε οι κυβερνήσει είναι ότι δεν υπάρχει πια τόσο μεγάλη επιδείνωση τη ανταγωνιστικότητα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και αυτό νομίζω πρέπει να το έχουμε υπόψη. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω, νομίζω αύριο λίγοι οι προθεσμοί για την κατάθεση τροπολογιών. Θα τι μελετήσω και αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι είμαι διατεθειμένο και να απαντήσω σε όλε τι τροπολογίε και να προσπαθήσω να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση όλοι εμείς οι οποίοι ε, μπλεκόμαστε σε αυτό το θέμα στο δυνατόν πιο αρμονικά. Ευχαριστώ. Grazie al relatore, ricordo che όπως ε, είπαμε, αύριο λίγη προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών και στις 24 Ιανουαρίου θα γίνει ψηφοφορία στην Ήτρα. Να σας υπενθυμίσω πριν ξεκινήσουμε την συνάντηση των συντονιστών ότι αύριο στις 9 είμαστε τις προσκεκλημένοι στην ε, ε, Επιτροπή Μεταφορών που είναι σε μια άλλη αίθουσα στο Γιάννα ε, Γιάν 4Q1 για να συζητήσουμε για τη χρηματοδοτική διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Στην 10 η ώρα όμως συνεχίζουμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Λοιπόν, σας ε, ζητώ τώρα να, αφήσετε, να εγκαταλείψετε την αίθουσα και να παραμείνουν εντός αιθούσης μόνο οι συντονιστές για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Bon.